good morning, Καλημέρα, συνάδελφοι. Ξεκινάμε τη σημερινή συνεδρίαση. Το πρώτο θέμα στην ημερήσια διάταξη σήμερα είναι το σημείο 7. Συμπερίληψη των εκπομπών αερίων θερμοκηπίου και των ε, απορροφήσεων από τη χρήση γης, ε, δασοκομεία κτλ. Και Δίνω τον λόγο στον κύριο Νόρμπερτ Λίντς. Ε, ευχαριστώ πάρα πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ για το ότι σήμερα συζητάμε αυτή την έκθεση, κυρίως της τροπολογίες. Έχουμε λοιπόν 15 τροπολογίες που είχα συντάξει εγώ προς την πρόταση της Κομισιόν και οι συναδελφοί συνολικά υπέβαλαν 277 τροπολογίες και βεβαίως υπήρχαν κάποια σημεία στα οποία δόθηκε ιδιαίτερο βάρος τα οποία θα ήθελα να αναφέρω συντομία ιδιαίτερα το βασικό θέμα του υπολογισμού του επίπεδου αναφοράς όπου είχαμε πολλές ε, τροπολογίες για τον υπολογισμό αυτών το χρονικό πλαίσιο αναφοράς πώς θα γίνει η αναθεώρηση τι ρόλο θα παίζει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη-μέλη και ε, βεβαίως το θέμα του πλαφών και αν θα πρέπει να υπάρχει πλαφών. πούμε παραδείγματος χάρη στην αναθεώρηση οι τροπολογίες κειμένονται από τροπολογίες που απλά προβλέπουν για την Κομισιόν έναν ρόλο τεχνικής υποστήριξης μέχρι ε, μία νέα μέχρι την Επιτροπή Δεσοκομείας, άλλοι ζητούν νέο υπολογισμό από τα κράτη-μέλη, εν μέρη υπό την Κομισιόν. είτε μια μεικτή επιτροπή με την Κομισιόν μέχρι προτάσεις που φτάνουν στο λεγόμενο net-net accounting ε, που λένε δηλαδή ότι ε, θα πρέπει ναι, όταν κόβεται δάσο να υπάρχει χρέωση, όπως λέγεται, ε, και όταν φυτεύεται δάσος να υπάρχει πίστοση. Για το χρονικό πλαίσιο αναφοράς μετά υπάρχουν προτάσεις ε, παράλληλα με αυτές τις κομισιόν που προέβλεπε από το 1999 μέχρι το 2009. Είχαν προτάσεις από το 2000 μέχρι το 2009, άλλοι λένε από το 2005 μέχρι σήμερα, άλλοι μέχρι το 2017, άλλοι προτείνουν να μην υπάρξει πλαίσιο αναφοράς. Το ίδιο και για το θέμα του αν θα πρέπει να υπάρχει πλαφόν, δηλαδή ποιες εκπομπές ή ποιο ποσοστό των εκπομπών θα υπολογίζεται στην δασοκομεία. Η Κομισιόν προτείνει 3,5% εγώ πρότεινα 7%. Υπάρχουν διαφορετικές τροπολογίες, άλλοι προτείνουν αύξηση για κάποια είδη ξύλου είναι να παραμείνουμε στο 3,5% και κάποιοι προτείνουν μια ομάδα προτείνει να υπάρξουν πολιτικά μέτρα για τον υπολογισμό των τιμών αναφοράς. Βλέπουμε λοιπόν ότι υπάρχουν μεγάλες διαφορές και Οπωσδήποτε θα προσπαθήσω ειδικά σε αυτά τα βασικά σημεία να προτείνω συμβιβασμούς και οπωσδήποτε θεωρώ πως αυτό το οποίο προτείνω εγώ βρίσκεται κάπου στο κέντρο των διαφόρων προτάσεων. Το επόμενο θέμα αφορά τα Harvest Good Products, τα λεγόμενα τα προϊόντα ξυλίας, δηλαδή μια α, ξεχωριστή κατηγορία προτείνουν κάποιοι συνάδελφοι πέρα από την πρόταση της Κομισιόν που λαμβάνει υπόψη ιδιαίτερα την ε, ξυλία κάποιοι συνάδελφοι ήθελαν να ληφθεί υπόψη η ιδιαίτερη εφορία του ξύλου ε, για το θέμα τώρα της γεωργίας ε, και του των εδαφών ε, αναφέρθηκε ιδιαίτερα το θέμα του πώς θα πρέπει ακριβώς από τώρα ήδη να δούμε και να αξιολογήσουμε τα υφιστάμενα περιβαλλοντικά μέτρα στο πλαίσιο του Λουλουσιεφ ε, που είναι το βασικό θέμα στην Γεωργία. Μετά υπήρχε η συζήτηση για τους υγροτόπους, αν θα πρέπει να περιληφθούν ή όχι. Και υπήρχε και εδώ πέρα κάποιες τροπολογίες ε, για την κατανομή των βαρών και την συζήτηση για την υποχρεωτική ή μη περίληψη των υγροτόπων ε, στο Λουρουσιεφ ε, και όχι στον κανονισμό για την κατανομή των βαρών και τελικά νομίζω ότι καταλήξαμε σε θα καταλήξουμε σε ένα αποτέλεσμα. Και τέλος, επειδή υπήρχαν πολλές τροπολογίες για την αναθεώρηση του κανονισμού, να υπενθυμίσω ότι και εκεί πρέπει να υπάρξει μια σύνδεση για και με την κατανομή των βαρών αλλά και με την Ενεργειακή Ένωση. Πρέπει να υπάρχει δηλαδή μια συνοχή όταν θα δούμε το τι θα γίνει μετά την πρώτη αναθεώρηση της Συμφωνίας των Παρισίων μετά το 2018 στο πλαίσιο του Λουλουσιεφ ε, και της ε, κατανομής των παρών. Είναι λοιπόν σημαντικό να βρούμε μια συνολική λύση. Αυτό αφορά λοιπόν ολόκληρο το κοινοβούλιο και βεβαίω κυρίω την έκθεση του συναδέλφου του κυρίου ε, Γκέρι Μπράντι. Αυτά ε, ω εισαγωγή από εμένα και αναμένω βεβαίω και το τι θα πούν οι συνάδελφοι. Thank you very much. And now we uh, Ευχαριστώ. Πάμε στους για τους φεστές πρώτα. Πρώτα ευχαριστώ. Όπως είπε ο συνάδελφος, υπάρχουν διάφορες ε, αποκλήσεις που ανέκυψαν εδώ. Όταν υπάρχει τόσο πάντων γιατί ομοφωνία, τότε υποχρεωτικά να ζητάς τις διαφορές. Η περίοδος αναφοράς νομίζω είναι συγκεκριμένη, μάλλον είναι ενδιαφέρουσα και θα πρέπει να το συζητήσουμε. Αλλά περιμένω κάποιον εδώ να τελειώσει τη συζήτησή του στο τηλέφωνο. Και υπάρχει και διάδρομο που να θέλετε να βγείτε. Η περίοδο του πάντων υπολογισμού είναι σημαντικό και ενδιαφέρον να εξεταστεί προσεκτικά ώστε να μπορεί ο καθένας να καταλαβαίνει τι γίνεται και ένα παράδειγμα που δίνω εδώ είναι το αν θέλει κανείς να κάνει δίαιτα για να μειώσει το βάρος του το προφανές θα ήταν να συγκρίνει το βάρος του το παρόν και το παρελθόν. Δεν έχει νόημα κανείς να κάνει δίαιτα αν συγκρίνει το βάρος του σε έξι μήνες. Γιατί μπορεί έτσι να κλέψει στο ζύγι. Αν λοιπόν το επίπεδο αναφοράς καθορίζεται για το μέλλον, αν η διαιτά σας τέλο πάντων καθορίζεται σχέση με το μελλοντικό σας βάρος, τότε το θα μπορείτε να κάνετε είναι να αποκτήσετε πολύ βάρος το επόμενο χρόνο, μετά να κάνετε δίαιτα και μετά να συγκρίνετε τον εαυτό σας έτσι, με αυτή την ε, εμφάνιση, με την εικόνα της ταχείας μείωσης βάρους. Οπότε αυτό δεν έχει νόημα. Και εγώ αναφορώ, ανα, συγγνώμη, ανησυχώ ότι αν η περίοδος αυτή καθοριστεί για το μέλλον και αν μια χώρα αποφασίσει ότι τέλο πάντων έχουν κομπεί πολλά δέντρα για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, τότε θα μπορούσε κάλλιστα να το συγκρίνει αυτό, να το αντιπαραθέσει τέλο πάντων με την μελλοντική περίοδο που θα έχει λιγότερε κοπέ δέντρων. Οπότε θεωρώ ότι η αναφορά θα πρέπει οπωσδήποτε να γίνεται στο παρελθόν και όχι στο μέλλον, γιατί αυτό ανοίγει αυτή λοιπόν η πρόταση της Κομισιόν αφορά κυρίως μια διαδικασία υπολογισμού ώστε τέλος πάντων να έχουμε ένα benchmark και να δούμε στην Ευρώπη τι γίνεται ακριβώ ώστε να κάνουμε συγκρίσει. Εγώ δεν έχω πρόβλημα οι αντιρρήσει σε σχέση με χώρε οι οποίε τέλο πάντων κόβουν πολλά δέντρα και τα χρησιμοποιούν, ιδιαίτερα σκανδιναβικέ χώρε έχουν θαυμάσιους πόρους και τους χρησιμοποιούν, τους αξιοποιούν. Αν όμως αποφασίσετε να κόψετε πάνω από την ετήσια σας αύξηση, τότε τίθεται κάποια ερωτήματα κατά πόσο έχει νόημα να κάνει κανείς κάτι τέτοιο, λόγω και κλιματικής αλλαγής. Αν κάποιος λοιπόν χρησιμοποιεί 80-85% της ετήσιας αύξησής του, τότε το ερώτημα, πέρα από το αν είναι καλό ή κακό, το ερώτημα είναι ότι τι γίνεται με αυτά τα δέντρα όταν κόβονται. Τι γίνεται λοιπόν αν όλες οι αιτήσεις αυτής σας χρησιμοποιούνται για, να, για την καύση, για παραγωγή ενέργειας. Η παραγωγή ενέργειας ας πούμε όταν γίνεται μέσω ξυλίας, εντάξει. Αλλά υπάρχουν χώρες οι οποίες χρησιμοποιούν μόνο 5-10% της ετησίας αύξησής τους. Και πρέπει να ρωτήσουμε του υπόλοιπου γιατί χρησιμοποιείται αυτό το θαυμάσιο πόρο τη στιγμή που θα πρέπει να καταπολεμήσουμε την κλιματική αλλαγή. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι κάνουν και άλλε χώρε και μετά να ρωτήσουμε ερωτήσει. Και όταν έχουμε ευρεία χρήση ξυλία, να δούμε τι γίνεται με αυτή την ξυλία, πώ χρησιμοποιείται. Αυτό θα πρέπει να ρωτήσουμε. Όχι απλά και μόνο σταθούμε στο γεγονό ότι χρησιμοποιούν πάρα πολύ την ξυλία. Ευχαριστώ. Βυσνιέσκα από το ομιλητής. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφοι, στη συζήτησή μας πολύ συχνά λέμε θα πρέπει να δράμε σφαιρικά, παγκόσμια. Και αυτό είναι σωστό. Αν θέλουμε πραγματικά να κάνουμε οι προσπάθειές μας να είναι αποτελεσματικές όσον αφορά την καταπολέμηση του διοξιδίου του άνθρακα, και τον ακουμπό του στην ατμόσφαιρα, τότε θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μα το παγκόσμιο πλαίσιο. Ξέρουμε ότι η Ένωση ευθύνεται για το 10% εκπομπή διοξιδίου παγκοσμίω. Έχουμε και τη Συμφωνία του Παρισιού που κατέστη δυνατή για ένα και μόνο λόγο ότι δεν περιλάβαμε την απαθρακοποίηση στο τελευταίο σχέδιο συμφωνίας και δεν αναφέρεται η μείωση διοξιδίου άνθρακα ως η μοναδική μέθοδος δηλαδή μείωση της μεγάλη συγκέντρωση διοξιδίου στην ατμόσφαιρα. Για τα υπόλοιπα η συμφωνία είναι σχετικά ουδέτερη όσον αφορά τις εκπομπές ρήπων. Εξάλλου έχουμε και θέματα όπως τα μέτρα απορρόφωσης, που έχουμε στα δάση μας, Οπότε, αν θέλουμε να τηρήσουμε το πνεύμα των Παρισίων, θα πρέπει να προωθήσουμε πολιτικές που θα αναπτύσσουν τα δάση μας και θα μας επιτρέπουν να τα διαχειριστούμε υπεύθυνα. Δυστυχώς, οι προτάσεις της Κομισιόν σε σχέση με το LULUCF απέχουν πολύ από αυτό. Για το LULUCF, λοιπόν, η έκθεση του κ. Λίντς κάνει κάποιες προσπάθειες, αλλά στις δικές μου τις τροπολογίες προτείνω να πάμε παραπέρα. Νομίζω θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας αυτά που γίνονται για την διαχείριση των δασών. Να θυμόμαστε επίσης ότι υπάρχουν κάποιες πρακτικές οι οποίε είναι αποτελεσματικές όσον αφορά το περιβάλλον. Επίσης θεωρώ ότι θα πρέπει να αφαιρέσουμε το 3,5% ως όριο όταν δηλαδή έχουμε να κάνουμε με, την, με ενσωμάτωση αυτών των προσπαθειών που γίνονται και θα πρέπει να αυξήσουμε αντίθετα το όριο όταν ε, έχουμε κάνει το Λολουσιεφ από τα 290 σε 425 εκατομμύρια. Και εδώ θα ήθελα να αφήσω την προσοχή σας στο γεγονός ότι ο τομέας δασοκομείας παίζει ένα πολύ σημαντικό ρόλο σε κάποιες χώρες όπως η Πολωνία όπου η κατάσταση εκεί είναι ιδιαίτερα σημαντική γιατί η μεγάλη πλειοψηφία των δασών ανήκουν στο κράτος. Τα περισσότερα δάση λοιπόν είναι κρατική περιουσία και έχουμε κρατικές επιχειρήσεις. Αν λοιπόν κάνουμε σωστές, ε, χαράξουμε σωστές πολιτικές, θα επιτρέψουμε και σε αυτές τις κρατικές υπηρεσίες να εφαρμόσουν σωστά τα μέτρα. Νομίζω ότι στην υπόλοιπη Ένωση βέβαια η διαχείριση των δασών είναι κάπως κατακαιρματισμένη, αλλά στην Πολωνία υπάρχει διαφορετική κατάσταση και ελπίζω η νέα πολιτική να λάβει υπόψη της ακριβώς αυτή την κατάσταση. Μετά στις τροπολογίες μου προσπαθώ να πετύχω μία συνέπεια μεταξύ τοπικών και πανευρωπαϊκών πολιτικών. Γιατί θεωρώ ότι εδώ πέρα μέσω αυτών των πολιτικών θα πρέπει να υπάρχει κάποια θεσμική ισορροπία και αυτό είναι αρμοδιότητα των χωρών μελών όσον αφορά δηλαδή, την διαχείριση των δασών. Δηλαδή η Κομισιόν δεν μπορεί να επιβάλλει επίπεδα αναφορά όταν έχουμε να κάνουμε τη δασοκομεία. Ο ρόλο τη ε, Κομισιόν θα πρέπει να περιορίζεται στην τεχνική υποστήριξη, στη μεθοδολογική υποστήριξη και στον έλεγχο των χωρών μελών. Πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μα όλε αυτέ τι διαφορέ όσον αφορά τη δομή τη ιδιοκτησία. Σα έδωσα το παράδειγμα τη Πολωνία προηγουμένω και σε πολλές άλλες χώρες τα δάση είναι κρατική περιουσία. Επίσης θεωρώ ότι αυτά τα όρια αναφοράς θα πρέπει να βασίζονται στα πιο επικαιροποιημένα και αξιόπιστα στοιχεία. Αυτό είναι ένα στοιχείο κλειδί όσον αφορά τη διαχείριση των δασών. Θα πρέπει λοιπόν επίσης να πούμε ότι η διαχείριση θα πρέπει να βασίζεται στι πραγματικέ δραστηριότητε και όχι μόνο στα ιστορικά ή στατιστικά δεδομένα. Θα πρέπει επίσης να προσβλέπουμε σε ένα επίπεδο διαχείρισης ε, δασών το οποίο πραγματικά θα αξιοποιεί το εθνικό δυναμικό διαχείρισης των δασών. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ από την ομάδα των φιλελευθέρων κύριε Στόρμπαντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ευχαριστήσω επίσης τον εισηγητή και τους ε, συναδέλφους ε, που συνεργάστηκαν ε, για να προκύψουν πολλές τροπολογίες, πολύ ενδιαφέρουσες απόψεις στο πλαίσιο μιας περίπλοκης διαδικασίας. Εγώ ξαγρύπνησα διαβάζοντάς τες και έμαθα πολλά πράγματα. Αλλά πέρα από αυτά που έμαθα, θα ήθελα να μην ξεφύγουμε από το βασικό μας στόχο, τον προσαρχικό μας ε, στόχο, που είναι η κλιματική αλλαγή και η αντιμετώπιση αυτής. Υπάρχουν πολλές ενδείξεις προς αυτή την κατεύθυνση. Πρώτο και κύριο, πάρα πολλές ασυνέπειες. Αυτές οι ασυνέπειες οδηγούν ε, στο ότι η δασοκομεία θα γίνει μια υπολοιπόμενη κατηγορία. Έχουμε ακόμη επιδοτήσεις για τον άνθρακα, δεν τα καταφέρνουμε στην, εκπομπή, στην εμπορία εκπομπών αερίων ε, και δεν ε, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα των δασών. Αν δούμε κανείς τα έγγραφα, τα συμπληρωματικά του IPCC, βλέπουμε ότι η αύξηση της ξυλίας είναι κάτι το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό Δηλαδή δεν θεωρούμε ότι τα δάση ε, είναι, ε, αποτελούνται από δέντρα και ότι είναι βασικά γιατί υπάρχουν πάρκα. Τα, θεω, τα, τα θεωρούμε σημαντικά για την ξυλία. Νομίζω λοιπόν ότι αν θέλουμε να κάνουμε μια διαχείριση των δασών κατά αυτόν τον τρόπο, δεν έχουμε πάρει τη σωστή κατεύθυνση. Δεν θέλουμε την ίδια αποτελεσματικότητα ε, από τη γεωργία όσον αφορά την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής. Το να κάνουμε λοιπόν τα δάση να πληρώνουν για τις ανεπάρκειες άλλων πολιτικών είναι κάτι κάτι το οποίο κάποιον ε, ικανοποιεί, αλλά όχι εμένα. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό ε, η ε, εισαγωγή Ε, σφαιριδίων από τις Ηνωμένε Πολιτείε και τον Καναδά. Και το λέω αυτό κυρίως για το Ηνωμένο Βασίλειο, τις κάτω χώρες, το Βέλγιο και τη Γαλλία. Και φαίνεται ότι είναι ικανοποιημένοι με την κατάσταση αυτή ε, και ε, θεωρούν ότι έτσι θα αντιμετωπίσουν τα προβλήματα των δασών. Δεν θέλω να μπω σε πολλές λεπτομέρειες, ε, αλλά νομίζω ότι μπορώ να επικεντρωθώ σε δύο βασικά προβλήματα. Πρώτα, η περίοδος αναφοράς και το 3,5% ανώτατο όριο. Ε, πρώτα απ' όλα για το χρονοδιάγραμμα. Η πρώτη διαδικασία του Κιώτο που επέβαλε ε, υποβολή εκθέσεων έγινε το 2001 και είχαμε πει ότι η περίοδος αναφοράς ήταν από το 2008 στο 2012 ε, είχε δηλαδή ένα χρονικό ορίζοντα 7 ετών. Λόγω των στατιστικών ε, αβεβαιοτήτων, ε, το ανώτατο όριο του 3,5% εισήχθη και όλοι συμφωνούσαν ή σχεδόν συμφωνούσαν με την προσέγγιση αυτή. Για τη δεύτερη περίοδο έγιναν πολλές αλλαγές όσον αφορά τις παραμέτρους ε, των εκθέσεων για να μην ε, υπάρχουν πλέον ε, αβεβαιότητες, όμως η γενική προσέγγιση διατηρήθηκε. Μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει στροφή 180 μοιρών ε, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και προτείνει ένα χρονοδιάγραμμα που, που κοιτάζει πίσω, ε, κοιτάνε προς το μέλλον α, ε, για να πάνε προς τα πίσω, κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο, ε, ε μου φαίνεται περίεργο αλλά χαίρομαι που διαβάζουν George Orwell στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. πρέπει να εξηγήσω το εξή. Η προτίμηση του να κοιτάμε προ το μέλλον, κοιτώντα προ τα πίσω, ήταν ε, λόγω της μεγάλης χρήσης της βιομάζας που έγινε το 2001. Ε, στη σελίδα 40 έχετε μία καμπύλη, υπάρχει μία κόκκινη γραμμή που δείχνει κάτι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Υπάρχει μία απότομη αύξηση στην κόκκινη καμπύλη που δείχνει ότι μεγαλύτερη ποσότητα βιομάζας χρησιμοποιήθηκε από ό,τι στο παρελθόν. Και υπάρχει και μία μικρή ενδιαφέρουσα λεπτομέρεια σε αυτήν την καμπύλη και είναι, βρίσκεται στο ίδιο επίπεδο με το επίπεδο αναφοράς. Αλλά αν δει κανείς ε, την πραγματικότητα και δει τις στατιστικές δεν υπάρχει απότομη αύξηση. Κοιτάξτε, εγώ δημοσιογράφος ε, είμαι στη σκέψη ε, και, αν, και σκέφτομαι πάντα μήπως κάνει κάποιος κάτι λάθος ε, στο παρασκήνιο. δεν ξέρω κατά πόσο λοιπόν είναι σύμπτωση το γεγονός ότι η κόκκινη γραμμή και το περίοδο και περίοδος αναφοράς συμπίπτουν. Εγώ πιστεύω ότι επίτηδες η κόκκινη γραμμή παρουσιάζεται κατά τέτοιο τρόπο. Το μοντέλο που χρησιμοποιεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι καταφανώς λάθος και θα έπρεπε να είναι σε θέση να κάνει κάτι γι' αυτό. Όσον αφορά τώρα το όριο του 3,5%. Αν έχουμε ένα ισχυρό σύστημα υποβολή εκθέσεων και συμφωνώ απολύτω με τον Πόλο ότι χρειαζόμαστε ένα τέτοιου είδου ε, σύστημα λογιστικό, θα έπρεπε όμω να υπάρχει τότε το ανώτατο όριο, γιατί η ετήσια αύξηση για την οποία πολύ καλά τοποθετήθηκε θα είναι μεγαλύτερη από τι δικέ μα δυνατότητε να τη χρησιμοποιήσουμε. Και αυτό θα δημιουργήσει πρόβλημα όχι για όσου φυτεύουν δέντρα σε μικρά ε, δάση. Αυτό είναι ε, πολύ καλό, αλλά δεν είναι η ουσία του προβλήματος. Ε, και αυτό με οδηγεί σε κάτι άλλο το οποίο πιστεύω ότι θα έπρεπε να συζητήσουμε. Είναι πώς γίνεται η υποβολή εκθέσεων για τη διαχείριση των δασών. Για την ώρα δεν υπάρχουν ποιοτικά στοιχεία για το τι σημαίνει διαχείριση των δασών. Μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα πάντα και αυτό δεν αποδεκτό. Τουλάχιστον όχι σε μένα. Συγγνώμη, θα ολοκληρώσω τώρα. Έχω κατακρίνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ε, προβλήματα και στην υποβολή της έκθεσης αλλά και στις προτάσεις της. Κάθε φορά που ζητήσαμε πληροφορίες βέβαια από την Επιτροπή μας τις έδωσε και θα ήθελα πραγματικά να τους ευχαριστήσω ε, από καρδιάς ε, γι' αυτό. Και θα σας ενοχλήσουμε λίγο παραπάνω ζητώντας σας και άλλες πληροφορίες γιατί νομίζω ότι έχετε πολλή γνώση σχετικά με το θέμα αυτό αυτό και θα τη, χρειαστούμε. Όσον αφορά όμως την έκθεση αξιολόγησης, κάτι πολύ ενδιαφέρον διαπίστωσα. Είδα την πρώτη έκθεση αξιολόγησης από την πρώτη περίοδο. Εκεί έκαναν μία προβολή ε, του, της τιμής του πετρελαίου, πολύ υψηλή, γιατί αυτές τις στατιστικές είχαν. Στη δεύτερη έκθεση αξιολόγησης προσάρμοσαν τους πραγματικούς, τις πραγματικές τιμές ε, για τα ιστορικά αριθμητικά στοιχεία που αφορούν το πετρέλαιο, αλλά η προβολή για το μέλλον ε, βασίζεται πάλι στην πρώτη αξιολόγηση, ε, κάτι το οποίο εμένα μου φαίνεται μάλλον παράλογο. Αυτά. Σας ευχαριστώ πολύ. Αυτή ήταν η πρώτη μου ε, παρέμβαση. Ε, θα συνεχίσω να συνεργάζομαι βέβαια με τους υπόλοιπους και όδης εισηγητές και με τον εισηγητή τον ίδιο. Ευχαριστώ πάρα πολύ κύριε Τόρουαλς. Δεν έχω θέσει χρονικό όριο για τις παρεμβάσεις, γιατί κάποιοι από τους σκιώδους εισηγητές δεν είναι εδώ, αλλά θα ήθελα παρόλα αυτά να ζητήσω από όσους παίρνουν το λόγο να σέβονται το χρόνο των συναδέλφων τους στις επιτροπές. Θα πάρω κι εγώ το λόγο και πρέπει να είμαι ο πρώτος που θα σεβαστεί αυτό το χρονικό όριο. Είμαι ο σκιώδης εισηγητής για τους πράσινους για το θέμα αυτό. Θα ήθελα καταρχά να ευχαριστήσω τον εισηγητή γιατί είναι εξαιρετική η δουλειά του και μπορώ να συμφωνήσω ότι υπάρχουν πολλέ διαφορετικέ προσεγγίσει και πολλέ τροπολογίε ε, επί του κειμένου. Δεν θα είναι εύκολο να ε, βρει κανεί το συμβιβασμό μεταξύ όλων αυτών των τροπολογιών. Παρ' όλα αυτά πιστεύω ότι με σκληρή ε, δουλειά θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε κάτι που θα είναι αποδεκτό από τις περισσότερες πολιτικές ομάδες και κυρίως ε, για την κοινωνία και το περιβάλλον. Όσον αφορά τώρα τα συγκεκριμένα ζητήματα, εγώ πιστεύω και συμφωνώ με την κυρία Βυσνιεύσκα ότι πρέπει να καταλάβουμε τον κανονισμό ε, Λουλούσιεφ στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και τις μακροχρόνιες, ε, στο πλαίσιο των μακροχρόνιων δεσμεύσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για την κλιματική αλλαγή, της Ευρωπαϊκής Ένωσης μάλλον, και πρέπει επίσης ε, να δούμε ε, τον κανονισμό δεν είναι ένα ζήτημα ε, γραφειοκρατίας, ένας λογιστικός μηχανισμός. Πρέπει να δούμε πώς ε, οι εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και οι απορροφήσεις ε, ε, βρίσκονται σε ισορροπία και πώς αυτό μας βοηθά να τηρήσουμε τις δεσμεύσεις μας στο πλαίσιο της Συμφωνίας των Παρισίων και ε, της αντιμετώπισης της κλιματικής ε, αλλαγής. Χρειάζεται λοιπόν μια σωστή λογιστική, ένας λογιστικός μηχανισμός σωστός, ε, αν θέλει κανείς να είναι πολύ κοντά στην πραγματικότητα, τι συμβαίνει στην, στην ατμόσφαιρα. Χρειαζόμαστε net-net accounting. Ε, για να μπορέσουμε να επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε συμφωνήσει στο Παρίσι και στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Νομίζω λοιπόν ότι η λογιστική περίοδος και ο καθορισμός αυτής είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Συνήθως έχω επικρίσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όμως νομίζω ότι καλό είναι να μείνουμε στην αρχική πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την περίοδο αναφοράς. Δεν μπορούμε να υποστηρίξουμε την τροποποίηση όπως προτείνεται από τον εισηγητή κατά τη γνώμη μας. Επίσης είναι πολύ σημαντικό και αναφέρθηκε και από τον εισηγητή ότι το θέμα δεν αφορά μόνη, τα, μόνο τα δάση. Οι, βιο, οι βοσκότοποι είναι επίση πάρα πολύ σημαντικά. Ε, σημαντικοί πρέπει να του συμπεριλάβουμε με κάποιο τρόπο. Πρέπει να έχουμε μία ριζοσπαστική ε, προσέγγιση όσον αφορά τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα από τη γεωργική δραστηριότητα ε, και ε, από το φαινόμενο χρήση γης και άλλα χρήσης γης. Το πρώτο βασικό ε, ζήτημα είναι το θέμα της βιοπικιλότητας. Ε, γιατί ε, ένα μεγάλο μερίδιο της ευρωπαϊκής ε, βιοπικιλότητας βρίσκεται στα, στα δάση της Ευρώπης. Όταν μιλάμε για το Λουλουσιέφ, μιλάμε κυρίως για την ετήσια αύξηση και την, ε, το, το, την επιφάνεια της, ε, των δασωμένων εκτάσεων. Δεν είναι μόνο το θέμα της ετήσιας αύξησης, αλλά το θέμα της ποιότητας των δασών που πρέπει να υπάρχει. Πρέπει και αυτό λοιπόν να το λάβουμε υπόψη την ποιότητα λοιπόν των δασών μας ε, αν απλώς ε, φυτεύουμε ε, ε, δέντρα για ξυλία, αν θέλουμε απλώς ένα απόθεμα διοξιδίου του άνθρακα ή αν θέλουμε δάση με υψηλού επίπεδου βιοπικιλότητα. Το θέμα είναι επίσης τα προϊόντα ξυλίας. Εγώ δεν διαφωνώ καθόλου με αυτό και με αυτή την προσέγγιση, αλλά πιστεύω ότι θα έπρεπε να είναι διαφορετικό το λογιστικό σύστημα που θα αφορά αυτό το θέμα, γιατί είναι ασαφές πώς αυτά τα προϊόντα ε, ε πώς ακριβώς γίνεται η λογιστική τους ε, μεταχείριση, αν είναι απόθεμα του διοξιδίου του άνθρακα ε, ή αν το, το κατά πόσο το διοξίδιο του άνθρακα που εκλείεται πηγαίνει πίσω στην ατμόσφαιρα. Οι εκπομπές από την βιοενέργεια πρέπει επίσης ε, να λαμβάνονται υπόψη λογιστικός πλήρως. Συμφωνώ ε, ότι μας βοηθάει η βιοενέργεια να ε, τηρήσουμε τις υποχρεώσεις μας, όμως δεν ε, είναι ε, παραγωγή ενέργειας. Το LULUCF τώρα ε, προφανώς συνδυάζεται με άλλους κανονισμούς, με τον κανονισμό ESR και πιστεύω ότι θα πρέπει να χρησιμοποιήσουμε περιορισμένη ευελιξία προκειμένου για το LULUCF για να μην δημιουργήσουμε κενά μεταξύ των διαφόρων κανονισμών. Και τέλος, αυτό είναι η τελευταία μου παρατήρηση και ελπίζω ότι τήρησα το χρονικό μου ε, περιθώριο είναι η διαφάνεια των λογιστικών ε, κανόνων και ισχυροί ε, λογιστικοί κανόνες, κάτι το οποίο είναι εύκολο να το καταλάβουμε, που θα είναι συγκρίσιμο μεταξύ των διαφόρων κρατών μελών και δίνει μια σαφή εικόνα του τι συμβαίνει στα δάση στην Ευρώπη. Ευχαριστώ. Αυτή ήταν η δική μου συνεισφορά στη συζήτηση. Και επειδή δεν βλέπω άλλον σκιώδη ηγητή από την ΚΟΕ και από την EFDD, θα ήθελα να ε, δώσω το λόγο σε συναδέλφους από την ε, Επιτροπή ε, το λόγο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα ήθελα και εγώ βεβαίως να στηρίξω τα επιχειρήματα του κυρίου Τόρβαλτς και να υπενθυμίσω ότι οι πρώτερες επιδόσεις της γεωργίας από το 1990 όπου είχαμε μία μείωση κατά 24 τις 100 εκπομπών είναι πάρα πολύ σημαντικές και βεβαίως η Ευρωπαϊκή Δασοκομεία συνεισφέρει ενεργά στην προστασία του κλίματος και φοβάμαι όπως και ο εισηγητή μας πως ε, τα δάση θα πληρώσουν τα λάθη άλλων τομέων. Γνωρίζουμε ότι ούτε 70% ε, των δασών δεν ε, χρησιμοποιείται και μπορούμε έτσι να αποθηκεύσουμε πολύ Περισσότερες εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα. Για εμένα βεβαίως σημαντικό είναι να βρούμε έναν καλό συμβιβασμό στο πλαίσιο των τιμών αναφοράς που θα έχει διαφάνεια και θα έχει έναν ισότιμο υπολογισμό για όλα τα κράτη-μέλη και βεβαίως για εμένα σημαντικό είναι οι εκπομπε. διοξιδίου του ανθρακά να μην πάνε απλά σε άλλες ε, χώρες ε, δεν είναι ε, νομίζω αυτή η πρόθεση κανενός ε, και για μένα είναι επίσης αναγκαίο να μην υπάρξει επιπρόσθετο διοικητικό βάρος για τους κατόχους δασών, τους ιδιοκτήτες. Πρέπει να διατηρηθεί η εθνική αρμοδιότητα, δεν είναι δυνατόν μέσω ευρωπαϊκών κανονισμών να παρεμβαίνουμε τόσο πολύ στην δασοκομεία. Επίσης πρέπει, θεωρώ εγώ, ήδη αυτά τα οποία έχουν γίνει σε πολλά κράτη-μέλη, ε, προστασία υγροτόπων, βιοπικιλότητα, να συμπεριληφθούν στην βάση υπολογισμού για να έχουμε μια σωστή βάση και έναν λογικό συμβιβασμό. Τέλος, Νομίζω πως θα είναι δύσκολο εγχείρημα για όλους τους συμμετέχοντες. Ε, εγώ βεβαίως έχω κάπως διαφορετικές προτεραιότητες ε, στη Γεωργία, αλλά είμαστε διατεθειμένοι για συμβιβασμό. Παρ' όλα αυτά θεωρώ πως η δασοκομεία και η Γεωργία είναι το κλειδί για μια επιτυχή εφαρμογή του Λουλουσίου, για μια επιτυχή κλιματική πολιτική σε τελική ανάλυση. Και θα τα δείτε αυτά και στις τροπολογίες μας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, επειδή ζητάνε πολλοί συνάδελφοι τον λόγο, δύο λεπτά ο καθένας. Αγίουζο. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι σκιώδης για την Ήτρε. Οπότε τα σχόλιά μου αφορούν αυτή την Επιτροπή. Έχουμε λοιπόν διάφορες τροπολογίες πολύ διαφορετικές μεταξύ τους. Δύο πράγματα. Για την μόλυνση αυτών των περιοχών. Νομίζω θα πρέπει να υπάρχει επικουρικότητα. Επειδή πραγματικά οι συνθήκες διαφέρουν μεταξύ των χωρών, δηλαδή από το βορρά στο νότο της Ευρώπης. Τώρα για την μακροχρόνια στρατηγική και τις τροπολογίες που αφορούν τα κρατικά, τα εθνικά σχέδια μέχρι το 2070. Η πρόταση της Κομισιόν στην διακυβέρνηση για το ενεργειακό πακέτο περιλαμβάνει κάτι παρόμοιο. Οπότε νομίζω θα πρέπει να θυγραμιστούμε και εμείς με την πρόταση αυτή. Τώρα, για το δίκτυο Natura 2000. Βεβαίω θα συνεχίσουμε να το εφαρμόζουμε, όμως εδώ έχουμε διάφορες προτάσεις που αφορούν την κλιματική αλλαγή, οπότε θα πρέπει να τα περδεύουμε τα, τα δύο αυτά θέματα για τις δασικές γέες και των υπολογισμών τους. Προτείνει η Κομισιόν περίοδο 20 ετίας, ώστε να θεωρηθεί δηλαδή αυτή η δασική περιοχή δάσος. Λαμβάνοντας όμως υπόψη το γεγονό ότι η κλασική περίοδος είναι η 20 ετία και μετά από την 20 ετία η ανάπτυξη είναι πολύ πιο αργή, θα πρέπει να βρούμε ένα μέσο όρο Υπάρχουν προτάσεις για περισσότερα, λιγότερα έτη, αλλά νομίζω 30 έτη είναι μια λογική περίοδος που εξυπηρετεί όλους. Μετά, για την ευελιξία που πρέπει να υπάρχει. Ευελιξία πρέπει να υπάρχει βεβαίω, αλλά επίση θα πρέπει να μην υπάρχει ευελιξία όσον αφορά τι φυσικέ διαταραχέ. Δυστυχώ εμεί έχουμε πάρα πολλέ πυρκαγιέ δασικέ και αυτό θα πρέπει να το λάβουμε επίση υπόψη μα. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πολύ. Δεν θέλω να καταχραστώ του χρόνου που μου δώσατε. Ευχαριστώ. Very much. Ευχαριστώ πολύ. Μπετήρ. Hvala vam, gospodine predsjedniče. Ε, prema članku 8 prijedloga uredbe... Ευχαριστώ. Υπό το άρθρο 8, το νέο, η νέα περίοδος αναφοράς θα οριστεί βάσει της ε, τρέχουσας πρακτικής μέχρι τώρα για τα εθνικά δάση, βάση της κατηγορίας τους, ε, όπως έχουν καταγραφεί από το 1999. Όσον αφορά την Κροατία, αυτό είναι ένα μεγάλο πρόβλημα λόγω των πολέμων που είχαμε, γιατί μεταξύ του 1990 και του 2009, το αναφερόμαστε δηλαδή σε αυτή την περίοδο, ε, είναι προβληματικό ε, για μας. Είναι σαν να λέτε ότι ό,τι αποφασίζεται ε, το 2009 ότι θα, θα αναφερόμαστε σε μια περίοδο από το 2001 ως το 2030. Όμως εμείς είχαμε πόλεμο. Ο πόλεμος αυτός είχε συνέπειες. Κάποια από τα δάση χάθηκαν και σχετικές υποδομές επίσης και λόγω της κατάστασης αυτής ήταν πολύ λιγότερο εντατική η διαχείριση των δασών. Από, για την περίοδο αυτή λοιπόν, από το 90 έως το 2000, μόνο 60% ε, του σημερινού ποσού έχει χρησιμοποιηθεί. Η συσσόρευση ξύλου θα μπορούσε να έχει αντίκτυπο και στις μελλοντικέ ε, ε, περιόδους αναφορών από την περίοδο του 2001 δηλαδή μέχρι το 2030. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε να υπάρξει μία εξαίρεση για την Κροατία, να χρησιμοποιηθεί μία διαφορετική περίοδος αναφοράς ε, για λογιστική... την λογιστικό υπολογισμό, σαν για μια περίοδος δηλαδή κατά την οποία οι συνθήκες ήταν πιο φυσιολογικές. Νομίζω ότι πρέπει να λάβουμε περισσότερο υπόψη τις ιδιαιτερότητες των κρατών μελών. Αυτό δεν έγινε. Όσον αφορά την ευελιξία, ε, λόγω του μεριδίου της γεωργίας από το 2001 στο 2010, ε, εμείς ε, για μας δεν είναι αποδεκτό και θεωρούμε ότι δεν έχει, επαρκώς, ε, δεν έχει επεξηγηθεί επαρκώς στην μελέτη αξιολόγηση επιπτώσεων. Θα υποβάλω και σχετικές πληροφορι... Ε, τροπολογίες. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα συμφωνήσω με την κυρία Μιλέ. Ε, βεβαίως η γεωργία είναι και πρόβλημα, είναι και μέρος της λύσης και μέρος του προβλήματο και πρέπει να δούμε τι θα γίνει και με τις εκπομπές μεθανίου. Πρέπει να έχουμε μια ρεαλιστική αντιμετώπιση. Γιατί βεβαίω, αν μιλάμε μόνο για την αλλαγή χρήση γη. τα τελευταία χρόνια βλέπουμε την μετατροπή των σκοτόπων που έχει απελευθερώσει πάρα πολλέ εκπομπέ και υγροτόπους ε, και την χρήση που γίνεται σε αυτούς και έχει άλλα προβλήματα που υποτιμούνται κάπως στην έκθεση. Και πρέπει βεβαίως να δούμε και τις εκπομπές ε, βιοενέργειας. Αυτό το οποίο με εκνευρίζει είναι το ότι έχουμε πάρα πολλά παραθυράκια και ευελιξία δηλαδή τους στόχους μείωσης που τους υπολογίζει ο καθένας όπως ε, θέλει και θα καταλήξει τελικά στο ότι ε, πολλές χώρες δεν μπορούν να... δεν είναι υποχρεωμένες να μειώσουν τελικά τις εκπομπές τους. Δηλαδή, τι λένε, κάνω δασοκομεία για να μην μειώσω τις εκπομπές ε, στην... στις μεταφορές. Όχι, δεν πάει έτσι δεν είναι βιώσιμη η πολιτική. Πρέπει να διατηρήσουμε τους στόχους σε όλους τους κλάδους, όχι να αντισταθμίζει ο ένας τον άλλον. Για την χρήση της ξυλίας πρέπει να το βλέπουμε αυτό μακροπρόθεσμα. Δηλαδή αν χτίζουμε ένα ξύλινο σπίτι είναι κάτι το διαφορετικό. Μπορούμε να μιλήσουμε για μακροπρόθεσμη θεώρηση. Αν παράγουμε χαρτί δεν είναι το ίδιο. Πρέπει λοιπόν να κλείσουμε περισσότερα παραθυράκια και να είμαστε, όπως σας είπα, πολύ πιο φιλόδοξοι. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Λίζε. Ο Νόμπετ Λίντς ε, πράγματι υπέβαλε μια πολύ καλή έκθεση και έχουμε κάποιες τροπολογίες για να τις ενισχύσει. Θεωρώ ότι είναι σημαντικό να στείλουμε το μήνυμα ότι πρέπει να στηρίξουμε ακριβώς μία αϊφόρο δασοκομεία Και βεβαίως ε, δεν θα γίνει αυτό χωρίς την ε, συμβολή της Γεωργίας και αλλά από την άλλη δεν πρέπει να στείλουμε το μήνυμα ότι αν κάποιος κάνει κάτι στην δασοκομεία μπορεί να μελήσει τους άλλους κλάδους. Όχι. Πρέπει να τα ζυγίσουμε και αν ισχύει, γιατί βεβαίως το θέμα είναι διεθνές, πρέπει να προσέξουμε η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην ε, αποτελέσει λάθος υπόδειγμα. Έχουμε χώρες με πολλά δάση, με λίγα δάση στην Ευρωπαϊκή Ένωση, αλλά αν δούμε το τι γίνεται διεθνώς, π.χ. τη Βραζιλία, προφανώς έχει πολύ περισσότερο δάσος από ότι ολόκληρη η Ευρωπαϊκή Ένωση. Λοιπόν, Ε, τι σημαίνει αυτό, ότι μέχρι το 2050 η Βραζιλία μπορεί να μην κάνει τίποτα ε, στις εκπομπές ε, της βιομηχανίας ας πούμε και των μεταφορών γιατί έχει τόσο τεράστια δάση. Όχι, δεν είναι έτσι. Δεν θα επιτύχουμε έτσι τους παγκόσμιους στόχους μας. Να είμαστε λοιπόν ευέλικτοι αλλά να μην χάνουμε το γενικότερο πλαίσιο. Και θεωρώ ότι τελικά όλοι θα πρέπει να δείξουμε κάποια εμπιστοσύνη στον Όρμπετ Λίντς, ο οποίος έχει κάνει μια καλή πρόταση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Η κυρία Ανταλή. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να ξεκινήσω υποστηρίζοντας την θέση του Πολ Μπρέναν ε, για το θέμα αυτό γιατί σε γενικέ γραμμέ συμφωνώ μαζί του. Ότι πρόκειται δηλαδή για ένα σημαντικό πυλώνα του πλαισίου για το κλίμα και την ενέργεια του 2030 και του Λελουσιεφ και θα ήθελα να εστιάσω σε αυτό στη μικρή μου παρέμβαση, ότι είναι δηλαδή ένα τμήμα μόνο της νομοθεσίας Λελουσιεφ, αλλά αυτό το οποίο θα ήθελα να τονίσω είναι η ευελιξία όταν μιλάμε ακριβώς ε, για τον ε, κανονισμό αυτών Και επίσης είμαι και σκιώδης ηγήτρια στο θέμα του ESR. Και πρέπει ακριβώς να δούμε την σχέση μεταξύ του Λουλουσιεφ και της εμπορίας απομπών και να μην καταλήξουμε με μια ευελιξία που θα είναι τόσο μεγάλη ώστε θα δημιουργεί τεράστια παραθυράκια που θα απειλεί την αξιοπιστία και την εφορία του σχετικού κανονισμού. Γιατί τελικά αυτό το οποίο έχουμε είναι μια ευελιξία για να βοηθήσουμε όλα τα κράτη-μέλη να επιτύχουν τους στόχους που θέλουμε μέχρι το 2030. Και βεβαίως ε, να μην ε, ξεχνάμε ότι έχουμε στόχους να πετύχουμε μέχρι το 2030. Θα ήθελα λοιπόν να αναφερθώ στην αξιολόγηση αντικτύπων, όπου η Κομισιόν αναφέρει ότι στο καλύτερο σενάριο μόνο 74 εκατομμύρια άδειών θα χρειαστούν έτσι ώστε να αντισταθμιστούν τα πιθανά ελλείμματα. Αναφέρει επιπλέον ότι ακόμα και αν τα κράτη-μέλη δεν μειώσουν τις εκπομπέ. 19 ε, εκατομμύρια πιστώσεις ε, Λουλουσιεύ θα απαιτηθούν η Κομισιόν. Ε, προτείνει 2 εκατομμύρια. Τροπολογίες πηγαίνουν σε διαφορετικές κατευθύνσεις. Άλλοι λένε να μην δοθεί καμία άδεια μέχρι 425 Και εδώ πέρα θα ήθελα να τονίσω ότι ναι, συμφωνώ να βρούμε έναν συμβασμό, αλλά να μην ξεπεράσουμε κατά πολύ το αναγκαίο για να επιτύχουμε και τους στόχους για το κλίμα και βεβαίως να φροντίσουμε ο κανονισμός να επιτύχει τους στόχους μας μέχρι το 2030. Και τέλος έρχομαι εδώ πέρα στις πιστώσεις ε, για την δασοκομεία, γιατί θεωρούμε ότι το σύστημα αυτό υπολογισμού δεν είναι σαφές αυτή τη στιγμή και έχει οδηγήσει σε υπερβολικές πιστώσεις στα κράτη-μέλη και τώρα έχουμε την ευκαιρία να το αντιμετωπίσουμε αυτό. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος Ζιμπ έχει τώρα τον λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ατέλειωτο το θέμα αυτό. Το θέμα της αναθεώρησης και της αξιολόγησης είναι πραγματικά τελείωτο. Πάντα θα υπάρχει ένα κενό όσον αφορά τις συγκρίσεις μεταξύ των χορμελών και τις διάφορες εμπειρίες, τις παραδόσεις, τις δομές που υπάρχουν, τη χρήση του εδάφους σε διάφορες περιοχές. Ας πούμε στη χώρα μου, τα τελευταία χρόνια είδαμε να υπάρχει μεγάλη ανάπτυξη των δασικών περιοχών, κάτι το οποίο ήταν βέβαια θετικό. Έγιναν πολλές αναδασώσεις. Αλλά και εκεί βέβαια θα πρέπει να δούμε κατά πόσο ας πούμε, οι καλλιεργήσιμες γέες θα πρέπει και αυτές έτσι να σχετίζονται με την ανάπτυξη του δάσους ή όχι, δεν ξέρω. Πάντως θα πρέπει για όλες τις χώρες ε, μέλη να ισχύσει βέβαια μια περίοδος αναφοράς και υπολογισμού, όμως η δομή ιδιοκτησίας είναι διαφορετική από χώρα σε χώρα, όπως στην Πολωνία, όπου έχουμε μια κρατική αρχή και υπηρεσία διαχείρισης δασών και η οποία καλύπτει την πλειοψηφία των δασικών εκτάσεων στη χώρα μας. Έχουμε λοιπόν τελείως διαφορετικό τρόπο διαχείρισης των δασών, έχουμε τελείως διαφορετικές προτιμήσεις και εδώ και πολλά χρόνια δεν δούμε περισσότερη σημασία στο να υπάρχει δασική υγεία αντί για καλλιεργήσιμη γη. Και το θέμα το ξέρω καλά, επειδή αντιμετώπισα το θέμα της δασικής διαχείρισης στην επαγγελματική μου ζωή. Ξέρω λοιπόν ακριβώς τι γίνεται με τη δομή της ιδιοκτησίας στην Πολωνία και ξέρω ότι υπάρχουν πολλά οικονομικά επίσης χαρακτηριστικά τα οποία καθορίζουν το επιχειρηματικό κομμάτι της δασοκομείας. Ε, υπάρχει το θέμα βέβαια το ιδιωτικό δάσος, το θέμα του κέρδους από το ιδιωτικό δάσος, υπάρχουν κοινωνικά ζητήματα επίσης. Ξέρω ότι έχω μόνο δύο λεπτά στη θέση μου και στην ουσία σας τα λέω αυτά πλατιάζοντας, αλλά τέλος πάντων αυτό που δεν πρέπει επουδενή να παραβλέψουμε είναι το θέμα των εδαφών και το δυναμικό που παρουσιάζουν όσον αφορά ακριβώς την απορρόφηση του άνθρακα. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε τι γίνεται με τη δομή σχετικά με αυτό των περιοχών αυτών. Θα πρέπει να δούμε τι γίνεται με τη γεωργική παραγωγή, τι λοιπάσματα χρησιμοποιούνται ας πούμε, τι χημικά προϊόντα χρησιμοποιούνται και μετά να δούμε κατά πόσο αλλάζει και το έδαφο. διαδικασία βέβαια καταλαβαίνω που δεν είναι εύκολη, θα πρέπει να ληφθεί υπόψη διαχρονικά και μην και δύσκολο και ευαίσθητο το σημείο. Πάντω ευχαριστώ που με ακούσατε. Ευχαριστώ λέει και ο Πρόεδρο, ευχαριστώ για τη συμβολή σα. Φτάσαμε τώρα στο τέλος των τοποθετήσεων από τα μέλη της Επιτροπής. Θα δώσω το λόγο τώρα στην Εκτελεστική Επιτροπή στην Κομισιόν. Ευχαριστώ. Καλημέρα σας συνάδελφοι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτήν την πολύ χρήσιμη συζήτηση και για την ταχεία πρόοδο σε αυτό το θέμα που πραγματικά την εκτιμούμε όλος ιδιαιτέρως. Βλέπουμε ότι είστε θετικοί και επικοδομητικοί δεν είναι περίεργο για μας, δεν αποτελεί έκπληξη για μας ότι ένα σημείο ανησυχίας είναι οι κανόνες ε, για τη λογιστική αντιμετώπιση των δασών. Να πω μία ακόμη φορά ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή βλέπει πολύ καθαρά ότι η ενεργός διαχείριση των δασών είναι πολύ σημαντική από απόψεως ε, κλίματος, ε, θεωρούμε ότι μπορεί να αποτελεί θετική συνεισφορά όσον αφορά την υποκατάσταση της ε, βάσης των ορυκτών ε, και των ε, πρώτων υλών. Θέλουμε όμως να είμαστε σαφείς ως προς το πώς θα συμπεριληφθεί αυτός ο τομέας και όλοι οι άλλοι τομείς που αφορούν τη γη. Ε, στην όλη διαδικασία επειδή έχουμε λάβει μια εντολή μέσω της Συμφωνίας των Παρισίων και κάποιου, κάποιοι από τους κανόνες, πολλοί από τους κανόνες που έχουμε προτείνει ε, εμείς βασίζονται σε αυτά που έχουν συμπεριληφθεί στο πρωτόκολλο του Κιώτο και εφαρμόζονται ήδη από τα κράτη-μέλη. Πολλοί από τους κανόνες ε, δεν ε, τους ανέπτυξε, ούτε τους εφήβρε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά τα κράτη-μέλη. Και το βασικότερο σημείο είναι τα επίπεδα δασών των κρατών μελών που έχουν οριστεί κατόπιν ετήματος των κρατών μελών, ώστε να επιτρέψουν τα εθνικά ε, χαρακτηριστικά των δασών τους να ληφθούν υπόψη. Νομίζω ότι αυτό είναι πολύ σημαντικό. Να ε, επισημάνω επίσης ότι όπως είπαν ήδη κάποιοι ευρωβουλευτές, ε, η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν είναι το μοναδικό συμβαλόμενο μέρος ε, είναι και άλλες αναπτυσσόμενες χώρες που κάνουν την ίδια προσπάθεια στο πλαίσιο της διαδικασίας Red Plus και οι περισσότερες αναπτυσσόμενες χώρες το κάνουν αυτό βάσει net-net accounting, χρησιμοποιούν δηλαδή ιστορικές τιμές αναφοράς και δεν έχουν πολιτικές συγκεκριμένες. Ε, ε, καλό θα ήταν η Ευρωπαϊκή Ένωση να μην δώσει το κακό παράδειγμα. Ε, όσον αφορά τουλάχιστον τις πολιτικές ε, ε, με μέσα αναφοράς που θα είναι στο μέλλον. Αυτό δεν δίνει ένα καλό παράδειγμα και καλό θα είναι να μην δικαιολογήσει αυτό ε, τη συνέχιση της βιοοικονομίας, το zero rating δηλαδή, ε, της ε, βιοενέργειας υπό το σύστημα εμπορίας εκπομπών αερίων. Αυτό βέβαια σημαίνει ότι υπάρχουν και πολλά οικονομικά κίνητρα, πολύ ισχυρά στο πλαίσιο της βιοοικονομίας. Θεωρούμε λοιπόν ότι είναι πολύ σημαντικό οι εκπομπές που συνδέονται με την καύση της βιομάζας να ε, λαμβάνονται ε, ορθά υπόψη και αυτό γίνεται στο πλαίσιο του κανονισμού Λουλουσιεύ ε, Είναι σημαντικό προκειμένου να συνεχίσουμε με την πολιτική μας. Παρεμπιπτόντως, οι Ηνωμένε Πολιτείε από τις οποίες όντως εισάχουμε πολύ βιομάζα και ε, ξύλινα ε, σφαιρίδια, κάνει, ήδη, κάνουν ήδη πολύ μεγάλη προσπάθεια, έχουν ήδη αναγνωρίσει το ότι έχουν συμπεριληφθεί ε, στις υποχρεώσεις τους ε, όσον αφορά τα προϊόντα ξυλίας που λαμβάνουμε από τα δάση και χρησιμοποιούν και εκείνοι το net net accounting, δηλαδή τις ιστορικές ε, τιμές αναφοράς. Για την περίοδο αναφοράς έχουμε δύο στοιχεία, κάνουμε προβολή των προηγούμενων ή των τρεχουσών πρακτικών ε, ε, διαχειρήσεων δασών στο μέλλον και ως δεύτερο στοιχείο δίνουμε τη δυνατότητα βάσει των χαρακτηριστικών του, των δασών του, στα κράτη-μέλη να εκτιμήσουν το επίπεδο βιομάζας που θα είναι διαθέσιμο στο μέλλον. Ε, αυτό το έχουμε εμεί εξετάσει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το χρησιμοποιούμε για την παρεκβολή ε, της ε, τρέχουσας διαχείρισης των δασών στο μέλλον 10% περισσότερα προϊόντα ε, θα έχουμε από τα δάση χωρίς την παραγωγή επιπλέον εκπομπών που πρέπει να τις λάβουμε υπόψη και σε λογιστικό επίπεδο. Αυτό δείχνει ότι οι τιμές αναφοράς για τα δάση που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι ένα ευέλικτο εργαλείο το οποίο δίνει τη δυνατότητα αλλά δίνει και κίνητρα για ενεργό διαχείριση των δασών. Η ανάλυση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στο πλαίσιο τη μελέτη τη ε, αξιολόγηση επιπτώσεων βασίζεται και σε καταλόγους ε, ε, και στατιστικά στοιχεία που έχουμε λάβει από τα κράτη-μέλη. Δεν έχουμε φεύγει τίποτε από μόνοι μα. Ευχαριστώ όμω να σα παρέχουμε περαιτέρω επεξηγή σε σχέση με όλα αυτά τα στοιχεία. Για την αναθεώρηση τώρα των τιμών αναφορά των δασών, ε, Αυτά όλα υπάρχουν στο πρωτόκολλο του Κιώτο. Ε, στο μέλλον ε, θεωρούμε και προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ε, οργανώνει τη διαδικασία αυτή με σαφή και πλήρη συμμετοχή των κρατών μελών. Κατά τη γνώμη μας όμως είναι σημαντικό να υπάρχει διαφάνεια πλήρη σε σχέση με το πώς έχουν οριστεί αυτά τα επίπεδα δασών και να υπάρχει μια ε, ε, ε, συνεκτική συνεισφορά όλων των κρατών η πρόταση Λουλουσιεύ υποστηρίζει την ενεργό διαχείριση των δασών και επίσης είναι συμβατή με το στόχο της αντιμετώπισης κλιματικής αλλαγής. Ευχαριστώ πολύ που μου δώσατε το λόγο. Ευχαριστώ και εγώ, λέει ο Πρόεδρος. Θα ήθελα να δώσω το λόγο στον ε, κύριο Λίν, στον εισηγητή, να συνοψίσει. Ναι, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ τους ε, συναδέλφους ε, για όλες τις συνεισφορές τους. Ε, τα σημείωσα όλα και τώρα έχω μια καλύτερη αίσθηση για το τι είναι σημαντικό για τις ε, τροπολογίες σας και το λάβω υπόψη όταν θα προσπαθήσω να γράψω συμβαστικές τροπολογίες ε, που θα συζητήσουμε σε 9 Μαΐου με τους να ε, Έχω προβλέψει τρεις τέτοιες συναντήσεις. Να δούμε αν θα φτάσουμε. Γιατί έχουμε και φιλόδοξο πρόγραμμα. Γεγονός είναι, το είδαμε και στην συζήτηση, πως ε, σε κάποια λεπτομερή ε, ζητήματα έχουμε μεγάλες αποστάσεις αλλά είναι σημαντικό αυτό το οποίο είπε και ο κύριος Πέτερ Λίζη, ότι καμιά φορά τίνουμε να βλέπουμε το δέντρο και να χάνουμε το δάσος. Και έχω την εντύπωση με πολλούς ομιλητές πως ε, δεν έχουν υπόψη τους ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρώτα απ' όλα πρέπει να διατηρήσει έναν ε, πρωτοποριακό ρόλο στα ζητήματα κλίματος και το ζήτημα είναι τι ε, διεθνείς ε, επιπτώσεις θα έχει κάτι τέτοιο. Αναφέρθηκε το παράδειγμα της Βραζιλίας. Τι επιπτώσεις λοιπόν θα έχει, η υψή απόφαση. Και γι' αυτό ακριβώς ελπίζω να τα συζητήσουμε και να βρούμε κάποιους συμβασμούς. Ε, κάτι ακόμα για τον κύριο Χόισλινγκ, ο οποίος ε, ανέφερε τον προβληματικό ρόλο της γεωργίας και δασοκομείας. Ε, πρέπει ακριβώς να τονίσουμε τον θετικό ρόλο, νομίζω, γεωργίας και δασοκομείας. Οπότε να δούμε και το τι έχει γίνει ιστορικά βεβαίως και ότι έχει συνεισφέρει η γεωργία αλλά ακριβώς να δώσουμε και ένα κίνητρο για να συνεχιστεί αυτός ο θετικός ρόλος. Και αυτό το οποίο ανέφεραν και άλλοι συνάδελφοι, δεν είναι δυνατόν η δασοκομεία να είναι δικαιολογία για να μην κάνουμε τίποτα σε άλλους τομείς. Ε, Ακριβώς όπως και άλλοι συνάδελφοι είπα και εγώ ότι όταν μιλάμε για ευελιξία και ε, βεβαίως είναι ένα ζήτημα του τι βαθμό πρέπει να έχει αυτή η ευελιξία ε, και είναι όμως απαραίτητη για την γεωργία και την δασοκομεία θα ήταν άσχημο όπως είπα να σημαίνει αυτό ότι θα έχουν έτσι μια επιταγή εν λευκό ή άλλη κλάδι. Σας ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Και για το χρονοδιάγραμμα τώρα θα ψηφίσουμε 22 Ιουνίου στην Επιτροπή και στην Ολομέλεια τον Ιούλιο. Τώρα θα δώσω την Προεδρία στην συνάδελφο, την κυρία Σάρμπου. Let's continue uh, with the exchange of views. Ας συνεχίσουμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με την έκθεση όσον αφορά την αποτελεσματικότητα της σύστασης 2014-70 για τις ελάχιστες αρχές για την έρευνα και παραγωγή υδρογών ανθράκων όπως το σχιστολιθικό αέριο με την, με την χρήση υδρορογμάτωσης μεγάλου, όπου τον λόγο έχει ο εκπρόσωπος ο κύριος Σαντάουσκας. Ελπίζω να είπα σωστά το ονοματάκι σας. Παρακαλώ. Ναι, ναι κύριε Πρόεδρε, μια χαρά. Κυρίε και κύριοι, κύριε Πρόεδρε, στις 14 Ιανουαρίου 2014 Κομισιόν ενέκρινε μια ανακοίνωση και σύσταση προς τα κράτη-μέλη για το σχιστολιθικό αέριο με κάποιες κοινέ αρχές για να υπάρχουν κάποιες δικλείδες ασφαλείας για το περιβάλλον και την υγεία κατά την εξόριξη σχιστολιθικού αερίου. Συγκεκριμένα τονίζουμε την ανάγκη προσεκτικού σχεδιασμού και επιλογής του τόπου υδρογραμμάτωσης, αξιολόγησης κινδύνου πριν ξεκινήσει η δρομάτωση, παρακολούθηση της ποιότητας των υδάτων και πληροφόρηση του κοινού. Η σύσταση συμπληρώνει την υφιστάμενη νομοθεσία που αφορά έργα που περιλαμβάνουν υδρορογμάτωση, όπως παραδείγματος χάρη την ε, αξιολόγηση δικτύπου ή την διαχείριση υδάτων ε, και απορριμμάτων. Και βεβαίως ε, αυτό είχε γίνει όταν αναπτυσσόταν ραγδαία στις ΗΠΑ η τεχνολογία αυτή, η εξέλιξη αυτή βεβαίως οδήγησε κάποιες προσδοκίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ένωση δηλαδή θα μπορούσε να ωφεληθεί και εκείνη και να έχει πρόσβαση σε νέες πηγές φυσικού αερίου και αργού πετρελαίου. Ε, δεν ε, επαληθεύτηκαν αυτές οι προσδοκίες. Ε, φαίνεται πως το κόστος παραγωγής στην Ευρώπη θα είναι υψηλότερο από ό,τι στη ΣΥΠΑ και επιπλέον τα σχιστολιθικά πετρώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση έχουν άλλα χαρακτηριστικά από ό,τι στη ΣΥΠΑ και βεβαίως η εκεί τεχνολογίες δεν έχουν οδηγήσει σε ανάλογες ε, βιώσιμες τεχνολογίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Στην έκθεση του Δεκεμβρίου 2016 η Κομισιόν επανεξέτασε τον κανονισμό με στόχο να δούμε πρώτα απ' όλα την διαχείριση του περιβαλλοντικού κινδύνου, δεύτερον να υπάρξει νομική βεβαιότητα για τις επιχειρήσεις, τρίτον να ανταποκριθούμε σε ανησυχίε του κοινού και τέταρτον να λάβουμε υπόψη την τεχνολογική πρόοδο και τις τεχνικές πέρα από την υδρορογμάτωση μεγάλου όγκου. Επίσης, λαμβάνουμε υπόψη την σχετική περιβαλλοντική νομοθεσία. Τα συμπεράσματα της ε, αναθεώρησης αυτής πρέπει να ειδωθούν υπό το πρίσμα του εξαιρετικά χαμηλού όγκου τέτοιων δραστηριοτήτων στην Ευρώπη σήμερα, καμία γεώτρηση η οποία θα επέτρεπε κερδοφόρο εκμετάλλευση δεν έχει γίνει πέρα από κάποιες ε, διερευνητικές ε, γεωτρήσεις. Τα δύο συμπεράσματα λοιπόν είναι τα εξή Πρώτον, η σύσταση έχει εφαρμοστεί με διαφορετικό τρόπο στα κράτη-μέλη και μη ικανοποιητικό σε κάποια. Δεν μπορούμε ακόμα να ξέρουμε την αποτελεσματικότητα της σύστασης ε, για την διαχείριση κινδύνων. Δεύτερον, τα κράτη-μέλη διαφέρουν στην εφαρμογή κάποιων διατάξεων ενώ βεβαίως ε, υπάρχει ακριβώς το νομικό πλαίσιο, οπότε δεν γίνεται πλήρως, πλήρης εκμεταλλευσή του. Παρ' όλα αυτά θεωρούμε ότι αν εφαρμοστεί σωστά, η σύσταση μπορεί να είναι ένα χρήσιμο εργαλείο για την διαχείριση κινδύνων, για την ανάπτυξη υδρογονανθράκων, απαιτείται όμως μεγαλύτερη πρόοδος και βεβαίως μια σωστή και ενιαία εφαρμογή του περιβαλλοντικού κεκτημένου. Στην έκθεση της ε, αναθεώρησης, η Κομισιόν ενθαρρύνει τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν τις ε, σχετικές αρχές της σύστασης σε άλλες μορφές ε, εξερεύνησης και εξόρυξης, μεταξύ των οποίων και η ενισχυμένη ανάκτηση τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, καταλήξαμε σε τέσσερις στόχους πρώτον αύξηση της διαφάνειας και της παρακολούθησης και αυτό θα γίνει μέσω μιας ε, πλατφόρμας διαδικτυακής η οποία θα κάνει μια απογραφή και χάρτη ε, που θα αφορούν ακριβώς τις γεωτρήσεις αερίου και πετρελαίου που δεν έχουν την παραδοσιακή μορφή δεύτερον. Έχουμε την εφαρμογή των σχετικών ε, διατάξεων για να στηρίξουμε τα κράτη-μέλη και τρίτος στόχος είναι να δούμε τους περιβαλλοντικούς κινδύνους και αντικτύπους των εξορρυκτικών δραστηριοτήτων, κοιτώντας τις βέλτιστες πρακτικές. Και τέταρτος στόχος είναι να δούμε το ερευνητικό κενό για τον αντίκτυπο στην υγεία. Αυτό θα γίνει με υφιστάμενους μηχανισμούς όπως ορίζοντας 2020 και θα ζητήσουμε μια γνωμοδότηση από την Επιστημονική Επιτροπή για τους περιβαλλοντικούς και υγειονομικούς κινδύνους. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να δώσω τώρα το λόγο στους... Ε, Χωρίς Αμπάνο. And then my colleague, sorry. Ευχαριστώ. Είχαμε την ανακοίνωση λοιπόν της Κομισιόν που μιλούσε για το θέμα αυτό της ρογμάτωσης σε σχέση με τους υδρογονάνθρακες. Πρέπει όμω να πούμε τρία πράγματα. Καταρχά ότι κατά την άποψή μα δεν υπάρχουν επαρκέ πληροφορίε και διαφάνεια και σε πολλέ περιπτώσει έχουμε υποβάθμιση των περιβαλλοντικών προδιαγραφών. Υποχώρηση που αποβλέψει δύο πράγματα. Στην πιο εύκολη εξόριξη και στην παροχή κινήτρων προς τους επενδυτές και τις πολυεθνικές. Νομίζω ότι η σύσταση δεν επαρκεί. Και η ίδια η Κομισιόν, όπως μόλις ανέφερε, λέει ότι αν εφαρμόσουμε σωστά τη σύσταση, αυτή θα μπορούσε να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο για την εγχείρηση των κινδύνων κτλ. κτλ. Το οποίο σημαίνει ότι στην ουσία αποδέχεται ότι δεν είναι χρήσιμη αυτή η σύσταση και ότι στην ουσία η κάθε χώρα κάνει ό,τι γουστάρει. Τώρα, η επίπτωση αυτής της κατάστασης είναι ότι παραβλέπουμε ή καθυστερούμε την αντιμετώπιση σοβαρών προβλημάτων περιβαλλοντικών, ενεργειακών κτλ. Θεωρούμε επίσης ότι οι κρατικοί προπολογισμοί δεν πρέπει να κινητοποιούν ή να ευνοούν ενεργειακούς ιδιασμούς που θα βασίζονται στα ορυκτά καύσιμα. Θα πρέπει λοιπόν να πάμε επιγόντως προς μια οικονομία χαμηλού άνθρακα με αποφάσεις όπως αυτές που αφορούν τη μείωση των ρήπων και την πρόθεση των ΑΠΕ. Θα πρέπει λοιπόν να πούμε ότι η χρήση του fracking στα πλαίσια αυτής της κρίσης ενεργειακής προκαλεί μεγάλη ζημιά και καθυστέρηση όσον αφορά ιδιαίτερα την χρήση ανανεώσιμων πηγών και βλέπουμε ότι αυτή μάλιστα έχει σταματήσει να εξελίσσεται σε πολλά μέρη της Ευρώπης. Θα ζητούσα λοιπόν από την Κομισιόν να διευρύνει το διάλογο που κάνει και στους ΟΤΑ τοπικές και περιφερειακές αρχές, γιατί και εκεί υπάρχει μεγάλο πρόβλημα έλλειψης διαφάνειας και πληροφοριών. Ευχαριστώ. Uh, uh, uh, ευχαριστώ πολύ κυρία Ντάλη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ πολύ την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που μας παρουσίασε τις λεπτομέρειες αυτής της αναθεώρησης. Δεν θα μπω στις ανησυχίες που αναφέρατε παρά το γεγονός ότι είναι αρκετά ανησυχητικές ε, όσον αφορά την ερμηνεία των κρατών μελών σε σχέση με κάποιες διτάξεις. Θα ήθελα να αναφερθώ στα τέσσερα σημεία για τα οποία, ε, στα οποία αναφερθήκατε ε, λέγοντας ότι σε αυτά θα επικεντρωθείτε. Αξιέπαινες είναι αυτές οι πρωτοβουλίες, αλλά θα ήθελα να ξέρω λίγο περισσότερα για το πώς θα λειτουργήσουν στην πράξη και στην πραγματικότητα. Στην πραγματική ζωή είπατε ότι θέλετε να αυξήσετε την παρακολούθηση και την διαφάνεια, που κατά τη γνώμη μου είναι εξαιρετικά σημαντικό, ειδικότερα αν πρέπει κανείς ε, να ε, λάβει υπόψη μια πρόσβατη έρευνα του Ευρωβαρομέτρου που έλεγε ε, που, αναφορούσε, που αφορούσε την, ε, τις δυνατότητες εξόρυξης στολιφικού αερίου στην περιοχή των ερωτηθέντων ε, και πόσο το έχουν ακούσει. Μία μικρή μειονότητα θεωρεί ότι είναι επαρκώς ενημερωμένη για τις δυνατότητες αυτές. Πιο συγκεκριμένα, και μιλώ για τη διαφάνεια εν προκειμένου, τα κράτη-μέλη έχουν εντελώς διαφορετικές προσεγγίσεις. Το Ηνωμένο Βασίλειο και η Ρουμανία δίνουν περιβαλλοντικές άδειε, αλλά δεν υπάρχουν αυτέ οι άδειε στη Λιθουανία και στη Γερμανία. Ε, τι κοινέ προδιαγραφέ θα μπορέσουμε να επιβάλλουμε ώστε να έχουμε παρακολούθηση και διαφάνεια πράγματι. Δεύτερον, είπατε ότι θέλετε να ενισχύσετε την ενιαία και ομοιόμορφη εφαρμογή του κανονισμού. Αξιέπαινο επίση. Αν δει κανεί όμω τα κράτη-μέλη, στο Ενωμένο Βασίλειο τώρα ολοκληρώνει περιβαλλοντικές ε, αξιολογήσεις επιπτώσεων ε, για την υδρορογμάτωση και δίνει νέες άδειες, αλλά από την άλλη η Πολωνία για παράδειγμα δίνει άδειες ε, χωρίς τέτοιου είδους αξιολόγηση. Πρόκειται λοιπόν για εντελώς αποκλίνουσες προσεγγίσεις. Και για το τρίτο που αναφέρατε όσον αφορά την αξιολόγηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων, πάρα πολύ θετικό μία, ε, μία, μία ακόμη φορά. Όμως δεν θεωρούμε ότι γίνεται συστηματική αναφορά από τους φορείς εκμετάλλευσης προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και για μένα αυτό είναι, σημαίνει ότι είναι εξαιρετικά δύσκολο να γίνει οποιαδήποτε αξιολόγηση περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Πάρα πολύ καλό είναι αυτό που μας λέτε και πολύ σημαντικό, αλλά πολλές φορές ε, καταφέρνουμε πάρα πολύ λίγα Οπότε θα ήθελα να μάθω λίγο περισσότερα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή πώς θα εφαρμοστούν όλα αυτά που προτείνετε τα τέσσερα σημεία στην πράξη και ε, πώς θεωρείτε ότι μπορείτε ε, όντως να δημιουργήσετε προστιθέμενη αξία από την εφαρμογή αυτών των τεσσάρων σημείων. Ο κ. Πεντετσίνη. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θεωρούμε ότι αυτή η ανακοίνωση για το φράκινγκ είναι περιορισμένη, έχει περιορισμένο εύρος, όπως ήδη υπόθηκε, γιατί αφορά μόνο την εφαρμογή σε έξι χώρες μέλη. Η Κομισιόν μας είπε ότι το αποδέχεται αυτό, επειδή ούτως θα εφαρμοστεί ακόμα και στις έξι χώρες αυτές με ανομοιογενή τρόπο. Κάποιε χώρε λοιπόν εφετούν αυτή τη τεχνική, άλλε όχι, όπω η Γαλλία και από ό,τι φαίνεται και η Γαλλία. Γιατί στη χώρα μα, το Υπουργείο Οικονομική ανάπτυξη, αρνήθηκε την χρήση του φράκινγκ. Παρόλο που κάποιοι εμπειρογνώμονες ε, διεθνώς είπαν ότι δεν είναι συμβατή αυτή η χρήση, χρησιμοποιείται από τη δεκαετία των 90 στην ε, περιφερειά μου, την Τοσκάνη. Δηλαδή στην ουσία τι κάνουμε. Έχουμε ένα τεράστιο ρεύμα υδάτων το οποίο τροφοδοτεί όλη την Νότια Ιταλία και αυτό το τεράστιο ρεύμα υδάτων μολύνθηκε από του υδρογονάθρακες και αυτό το νερό αυτή τη στιγμή πίνεται από εκατομμύρια Ιταλούς πολίτες και αυτή είναι μια μάχη που δώσαμε εδώ και καιρό. Ένα από του λόγου αυτής τη μόλυνσης ήταν ακριβώ η χρήση του φράκινγκ σε αυτέ τι περιοχέ, εν αγνία του πληθυσμού. Πράγματι η έκθεση της Κομισιόν δεν αποκλείει το ενδεχόμενο η Ιταλία να εξαιρεθεί από το σύνολο των χωρών που θα εφαρμοστεί το φράκινγκ. Η Κομισιόν λέει επίση ότι η Ιταλία είναι μια από τι 11 χώρε οι οποίε επιβεβαιώσαν ότι προτίθενται να δώσουν άδειε για μη σημαντικού τύπου και σταθμού υδρογοναθράκων με υποβοηθούμενη ανάκτηση. Αν όμως δούμε τις εκθέσεις αυτές, θα καταλάβουμε ότι η Ιταλία λέει ότι ακριβώς για να βελτιώσει την ανάκτηση συγκεκριμένη παραγωγής μπορεί να χρησιμοποιηθούν τεχνι... τεχνικές που στην ουσία είναι το fracking. Οπότε το ερώτημα εδώ είναι, όταν η Ιταλία και άλλες χώρες λένε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι επιτρέπονται τεχνικές ε, όσον αφορά τους άνθρακες, δεν επιτρέπουμε αυτό τον τρόπο την χρήση τεχνικών οι οποίες στην ουσία είναι ρογματώσεις. Θα πρέπει λοιπόν να επιτρέπουμε τη ρογμάτωση όταν έχουμε να κάνουμε με σχιστολιθικό ή άλλου υδρογονάθρακες. Και τι γίνεται με το περιβάλλον σε αυτές τις περιπτώσεις και, τις, ε, και την κατάστασή του σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Η κυρία Ντονάνο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Αυτή η έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής επιβεβαιώνει τους κινδύνους που έχουν να ε, κάνουν με την υδρορογμάτωση όχι μόνο για την εκμετάλλευση του σχιστολιθικού αερίου αλλά και άλλων ορυκτών καυσίμων ε, μη συμβατικών ε, όπως και από τον άνθρακα για παράδειγμα. Στη Γαλλία υπάρχουν σημαντικοί τέτοιοι πόροι. Όταν όμως αυτοί οι πόροι βρίσκονται σε βάθος μικρότερο από το κοίτασμα, ε, η υδρορογμάτωση θα σήμαινε ότι ε, ο κίνδυνος ήταν ακόμη μεγαλύτερος. Ένας κίνδυνος ε, μόλυνσης του πόσιμου νερού, όπως επίσης υπάρχει περίπτωση μεγάλης, χρήσης μεγάλου όγκου υδάτων. Ε, α, επομένως πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει ε, ανάκτηση όλων αυτών των ε, κοιτασμάτων, όμως η έκθεση λέει ότι δεν υπάρχει καμία διαδικασία ε, που να μπορεί να ε, αντισταθμίσει τους κινδύνους, όπως για παράδειγμα η νανοτεχνολογία. Πρέπει να βρούμε νέους τρόπους εκμετάλλευσης που να σέβονται περισσότερο το περιβάλλον και αυτό θα έδινε τη δυνατότητα βελτίωσης του να λαμβάνεται υπόψη πρόοδος και, και οι νέες τεχνικές στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης όσον αφορά αφορά την παραγωγή τέτοιου είδους υδρογων ανθράκων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και εγώ. Ο κύριος Τέιλ. Yes, sorry, Chair. Thank you very much. Um... Ευχαριστώ πολύ. Νομίζω ότι το πρώτο σημαντικό που θα έλεγα είναι ότι πολλοί εξημών... Αχ, συγγνώμη, ξέχασα να κλείσω το κινητό μου. Uh, Πολλοί από εμά ανησυχούσαμε το 2014 όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε πάρα πολλές συστάσει και νομίζω ε, ότι το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε όπως επιβεβαιώνεται από την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ε, χάλια. Ε, σε πολλές περιπτώσεις ε, οι εταιρείες πετρελαίου και αερίου ουσιαστικά θέτουν τις ε, δικλίδες ασφαλείας περιβαλλοντικές που θεωρούν ότι είναι απαραίτητες εκείνες. Εμείς, αυτές όμως είναι εντελώς διαφορετικές από αυτές που πιστεύουμε εμείς ότι θα έπρεπε να υπάρχουν. Χρειάζεται ένας δεσμευτικός κανονισμός. Πιστεύω λοιπόν ότι θα έπρεπε, επαναλαμβάνω και συστήνω να υπάρξει ένας δεσμευτικός κανονισμός. Την περασμένη εβδομάδα ήταν εβδομάδα περιφερειών ε, και μιλούσαμε ε, πολλές ε, ε, πήγα σε πολλές ε, διερευνητικές εξορίξεις ε, πετρελαίου και σχισολιστικού αερίου στο Ηνωμένο Βασίλειο και βλέπουμε ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες. Βέβαια υπάρχει μεγάλος κίνδυνος μόλυνσης των υδάτων της ατμόσφαιρας. Έχω πάει στην Πενσιλβάνια, έχω δει τι αποτελέσματα υπάρχουν από τέτοιου είδους εκμετάλλευση. Είναι αρνητικός ο αντίκτυπος και για τον κόσμο και για το περιβάλλον τους. Τώρα, για να μπούμε στις λεπτομέρειες της έκθεσης, ε, συμφωνώ με τις ανησυχίες που έχουν αναφερθεί ε, και αλλού όσον αφορά τον ορισμό ε, της μεγάλου όγκου υδραυλικής ρογμάτωσης στη Νότια Αγγλία. Συμβαίνει τώρα συνεχώς, οι εταιρείε πετρελαίου και αερού να λένε όχι, δεν χρειάζεται να ανησυχείτε γιατί εμείς δεν κάνουμε υδρορογμάτωση. Εμείς απλώς χρησιμοποιούμε την ε, ενεργοποίηση του κοιτάσματος για να μπορέσουμε να πάρουμε ε, το πετρέλαιο και το αέριο. Όμως ε, η, η η κατάσταση αυτή είναι ένα είδους, ενός είδους ρογμάτωση, έχει το ίδιο αποτέλεσμα γιατί φτάνουμε μέχρι τον πάτο της πηγής και, δημιουργούμε πολύ μεγάλη πίεση για να δημιουργηθεί ρόγμα, ρογμή στο πέτρωμα και αυτό χρησιμοποιεί πολύ περισσότερο τοξικές χημικές ουσίες από την κανονική υδρορογμάτωση. Ε, γιατί το υγρό που χρησιμοποιείται κυρίως για την υδρορογμάτωση ε, είναι κυρίως νερό με 0,5 5% άλλες χημικές ουσίες, ενώ στην άλλη περίπτωση τα χημικά είναι ε, περίπου 18%. Αν λοιπόν προσπαθούμε να ε, μειώσουμε τον κίνδυνο και να είμαστε ασφαλείς, ε, τότε ο ενδεχόμενος κίνδυνος είναι κάτι που πρέπει να τον λάβουμε υπόψη. Πρέπει να διευρύνουμε τον ορισμό ε, ε, πολύ περισσότερο από αυτόν που προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ελπίζω, νομίζω, ελπίζω, ε, νομίζω επίσης ότι πρέπει να δώσουμε ιδιαίτερη σημασία στην υποβολή εκθέσεων περιβαλλοντικών και πιστεύω ότι πρέπει να ε, έχουμε ε, να, να, υδρορογμάτωση να γίνεται μακριά από ευαίσθητα μέρη ε, όπως ε, για παράδειγμα περιοχές όπου υπάρχουν μεγάλες ποσότητες νερούς, νερού, λίμνες για παράδειγμα και άλλου είδους περιβαλλοντικώς ευαίσθητα μέρη. Νομίζω ότι το πιο ε, σημαντικό που μπορούμε να κάνουμε είναι να μην έχουμε απλώς συστάσεις, αλλά ε, κανονισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Το είπαν οι συνάδελφοι. Το ερώτημα είναι τι θα γίνει από εδώ και μπρος. Και διαβάζω στην έκθεση της Κομισιόν. Έχει νομίζω κάποια συμπεράσματα τραγικά για το πώς εφαρμόζεται η περιβαλλοντική νομοθεσία στην Ένωση αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Και βεβαίως, ε, εντάξει, η Κομισιόν λέει διαφορετική ερμηνεία κάποιων διατάξεων της νομοθεσίας, αλλά αυτό το οποίο σημαίνει είναι ότι το νερό δεν προστατεύεται. Ότι οι χώρες δεν κάνουν τα όσα θα έπρεπε να κάνουν σύμφωνα με την οδηγία περί εξορρυκτικών δραστηριοτήτων, υδάτων ή εκπομπών. Είναι πολύ σκληρά συμπεράσματα και βεβαίως ε, ε, ποιο είναι η σύσταση, περισσότερος ε, διάλογος. Λοιπόν, προτείνω το εξής. Όταν κάνετε την αξιολόγηση το 2014 υπήρχαν τέσσερις πιθανότητες. Μία μη δεσμευτική σύσταση και οι άλλες τέσσερις ήταν πολύ σκληρότερες. Ε, ακόμα και πήγαιναν σε συγκεκριμένες, σε οδηγία η οποία θα κάλυπτε τα ζητήματα. Δηλαδή από πολύ γενικές συστάσεις μέχρι οδηγία. Τέσσερις επιλογές. Ενώ στην αξιολόγηση αντικτύπου η Κομισιόν γνωρίζει ότι αν θέμε να μιλάμε σοβαρά πρέπει να κάνουμε οδηγία αλλά επέλεξε μια μη δεσμευτική σύσταση. Τώρα, μετά από τρία χρόνια, ερχόμαστε και λέμε «Ε, οι μη δεσμευτικέ συστάσεις δεν κάνουν τίποτα. Και η σύσταση είναι α, και άλλος διάλογος. Ε, εγώ απορώ. Η ερώτησή μου λοιπόν είναι απλή. Οι τέσσερις αυτές επιλογές ε, του 2014 υφίστανται ακόμα? Εάν ναι, τι πρέπει να γίνει τα επόμενα χρόνια μέχρι να πάει προς αυτές τις επιλογές η Κομισιόν ή επιμένουμε στην επιλογή που ξέρουμε ήδη ότι δεν έχει αποτελέσματα. Αυτή είναι η ερώτησή μου. Ευχαριστώ. Κάποιος άλλος θα ήθελε να μιλήσει. Όχι. Θα δώσω λοιπόν το λόγο πάλι στην Κομισιόν να δούμε τι θα μας πει. Σας ευχαριστώ για αυτά τα οποία μας είπατε και για τα σχόλια. Να ξεκινήσω από το πλαίσιο. Το 2014 λήφθη κάποια δράση γιατί πολλοί θεωρούσαν ότι η εκμετάλλευση των μη συμβατικών πηγών θα απογειωνόταν. Κάτι το οποίο δεν συνέβη. Δεν έχουμε ούτε μία εμπορική εκμετάλλευση στην Ευρώπη. Τίποτα. Τίποτα. Έχουμε κάποιες εξαιρετικές γεωτρήσεις, αλλά δεν υπάρχει εμπορική δραστηριότητα. Δεν είμαστε όπως τις είπα. Αυτό λοιπόν πρέπει να το έχουμε υπόψη. Το έχουμε υπόψη το πλαίσιο ότι η κλίμακα της εκμετάλλευσης είναι ε, σχεδόν μηδενική. Και αυτό υπαγορεύει και την μορφή του μέσου που θα χρησιμοποιήσουμε. Ναι, γεγονό είναι ότι η σύσταση είναι ένα ήπιο μέσο, μπορείτε να πείτε, αλλά το ερώτημα είναι εάν αυτή τη στιγμή όταν ε, δεν υπάρχει εμπορική εκμετάλλευση αξίζει τον κόπο να κάνουμε άλλο ένα νομικό μέσο. Νομίζω ότι δεν θα είναι αναλογικό. Επιπλέον, μπορεί να αντιμετωπίζουμε το ίδιο πρόβλημα και με νομικά μέσα. Αν έχουμε οδηγία ή κανονισμό, μπορεί πάλι να έχουμε μη συμμόρφωση. Ναι, εντάξει, έχουμε κάποια άλλα μέσα επιβολής, αλλά αυτό δεν σημαίνει πάντα ότι εφαρμόζονται στην πράξη. Όχι πάντα. Μάλιστα, έχουμε μια περίπτωση ήδη ενώπιον του δικαστηρίου κατά ενός κράτους μέλους, ας πούμε το πιο ενεργό στον κλάδο αυτόν, ή το δεύτερο ίσως πιο ενεργό, λόγω μη συμμόρφωσης με την ε, αξιολόγηση περιβαλλοντικού αντικτύπου. Έχουμε λοιπόν κυρώσεις στην ομοθεσία για τα ζητήματα αυτά. Η σύσταση λέει απλά ποια νομοθεσία ισχύει για ποιος ε, υδρογονάνθρακες και πώς πρέπει να εφαρμοστεί. Έχουμε λοιπόν ένα νομικό κείμενο και εφαρμοστεί. Επίσης έχουμε την οδηγία ποσίμων υδάτων, ε, την οδηγία για τα εδάφη. Αυτά πρέπει να ισχύσουν και στις περιπτώσεις αυτές. Έχουμε λοιπόν νομικά κείμενα. Απλά πρέπει να εφαρμοστούν. Και αυτό είναι το πρόβλημα που βλέπουμε στην έκθεση και το λέμε ξεκάθαρα. Δημοσιεύσαμε επί τη ευκαιρία, νομίζω τη εβδομάδα που μας πέρασε, τις απαντήσεις των κρατών μελών. Ε, προς τις προς τα αιτήματα της Και αυτά πρέπει βεβαίως ε, να τα παρέχουν κάθε χρόνο τα κράτη-μέλη. 26 ακόμα απαντήσεις περιμένουμε. Αλλά νομίζω αυτό δείχνει την κλίμακα των δραστηριοτήτων που είναι χαμηλή θα έλεγα και νομίζω έτσι να απαντηθούν και κάποιες ε, ε, από τις απαιτήσεις διαφάνειας. Θα δούμε δηλαδή τι κάνουν τα κράτη-μέλη και έτσι θα μπορέσουμε να κρίνουμε το εάν ε, η ερμηνεία της ε, νομοθεσίας είναι αυτό το οποίο υποψιαζόμαστε ή αν δεν είναι τόσο προβληματική. Αλλά βεβαίως αυτό δεν ε, σημαίνει κάτι για τη διαφάνεια. Έχουμε προγραμματίσει λοιπόν κάποιες δράσεις. Η πρώτη για την διαφάνεια όπως σας είπα είναι ο διαδραστικός χάρτης και Εκεί θα θέλαμε να έχουμε ένα πιο χρήσιμο διαδραστικό μέσο και να ξέρουμε πού είναι η γεώτρηση, ποιες άδειες έχουν δοθεί, ποιος την εκμεταλλεύεται, τι ουσίες χρησιμοποιούνται και όλα αυτά. Αυτό θα θέλαμε να το δημοσιοποιήσουμε. Θα έχουμε την πρώτη δοκιμή, ελπίζουμε, δοκιμαστική έκδοση το καλοκαίρι και θα έχουμε και χρήσιμες πληροφορίες έτσι ώστε οι πολίτες και το κοινό να δουν το τι ε, συμβαίνει στον τομέα αυτόν. Για τον ορισμό τώρα της ε, ρογμάτωσης. γνωρίζουμε ότι η σύσταση ισχύει για τους υδρογονάνθρακες ε, και το σχιστολιθικό αέριο ιδιαίτερα. Έχουμε τον ορισμό του τι σημαίνει και στις περισσότερες περιπτώσεις σημαίνει η χρήση ε, νερού πράγματι αλλά υπάρχουν και χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται καμιά φορά και θα θέλαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα μέσα που έχουμε π.χ. τον κανονισμό REACH για να γνωρίζουμε τις ιδιότητες των χημικών ουσιών. Εάν ο κανονισμός είναι πολύ περιορισμένος, μπορεί να ισχύει κάτι τέτοιο, τουλάχιστον τότε περιμένουμε τα κράτη-μέλη να εφαρμόσουν το πνεύμα και όχι μόνο το γράμμα του κανονισμού. Γι' αυτό χρειάζεται διάλογος, να κάτσουμε με τα κράτη-μέλη και να δούμε πώς βλέπουν τις λεπτομέρειες ε, της σύστασης και αν χρειάζεται να αναθεωρηθεί κάτι. Υποσχεθήκαμε να το κάνουμε αυτό τακτικά, αλλά χρειαζόμαστε ακριβέστερες πληροφορίες για το τι συμβαίνει πριν υποσχεθούμε κάτι για νομοθετική ή μη νομοθετική δράση. Αλλά θα θέλαμε να εκμεταλλευτούμε όλες τις δυνατότητες που έχουμε τώρα. Να έχουμε διάλογο σωστό με τα κράτη-μέλη, να δούμε το τι μπορεί να γίνει, να δώσουμε στα κράτη-μέλη μια ευκαιρία μέσω κάποιων ερμηνευτικών κειμένων να εφαρμόσουν ε, σωστά την νομοθεσία και αν δεν γίνει κάτι τέτοιο να το ξαναδούμε. Αυτή είναι η απαντήση μου. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Περνάμε στο επόμενο σημείο. Ανταλλαγή απόψεων με την Επιτροπή σχετικά με το πρόγραμμα βελτίωσης ε, και αποδοτικότητα του ασφαλιστικού πλαισίου REFIT για το οικολογικό σήμα ΕΜΑΣ. Έχετε πάλι τον λόγο εσείς, η Κομισιόν. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Περίμενα να τελειώναμε σήμερα στη συνεδρίαση αυτή, δηλαδή την εξέταση των δύο θεμάτων. Αλλά δυστυχώς δεν είμαι σε θέση να πω ότι θα το κάνουμε γιατί είμαστε στην τελική φάση της έκθεσής μας για το ΕΜΑΣ και την οικοσήμανση. Ελπίζω πάντως να την ολοκληρώσουμε την έκθεσή μας ε, προσεχώς. Τώρα, για το σχέδιο δράσης κυκλικής οικονομίας. Αυτό ζητά από την Κομισιόν να ολοκληρώσει ακριβώ τον έλεγχο και η Κομισιόν τον έχει ξεκινήσει βέβαια και καταλαβαίνουμε και τι ανησυχίε των εμπλεκομένων σε σχέση με την καθυστέρηση τη υιοθέτηση των συμπερασμάτων του ελέγχου. Και ελπίζω το εξάμεινο αυτό το τρέχο να μπορέσουμε να ολοκληρώσουμε να ολοκληρώσουμε την αξιολόγηση αυτή που θα πρέπει να περιλαμβάνει δύο έγγραφα. που θα αφορούν λεπτομερείς τέλο πάντων αναλύσεις των υπέρ και των κατά επιτυχιών και αποτυχιών και μια έκθεση επίσης της Κομισιόν με κάποια σκέψη για το μέλλον. Θα ακολουθήσουμε πάντως τις παρουσιακές, ε, παρουσιακά πέντε κριτήρια σε αυτές τις περιπτώσεις, αποτελεσματικότητα δηλαδή, συνέπεια, συνοχή κτλ. Ήδη ξέρουμε από τώρα ότι ένα από τα προβλήματα που συχνά αντιμετωπίζουμε είναι η πρόσληψη. Η πρόσληψη η οποία είναι πολύ χαμηλή για αυτά τα εργαλεία ώστε να έχουν πραγματική επιρροή. Οπότε θα πρέπει να σκεφτούμε το πώς θα μπορούσαμε να προωθήσουμε αυτά τα δύο εργαλεία και να δούμε τι άλλο θα μπορούσαμε να κάνουμε ώστε τα εργαλεία αυτά να γίνουν πιο δημοφιλή μεταξύ των επιχειρήσεων και των δημοσίων αρχών. Οπότε αυτά υποχρεωτικά έχω να σας πω αρχικά, αλλά προτείνω να επανέλθουμε για το θέμα αυτό στην Επιτροπή σας όταν θα έχουμε περισσότερα αποτελέσματα και μετά από συζητήσεις με χώρες μέλη για να δούμε και αυτές πόσο έτσι θέλουν να προωθήσουν αυτά τα εργαλεία τα οποία θεωρούμε ότι έχουν μέλλον. Ευχαριστώ. η πρόεδρο, μήπως κάποιος θέλει το λόγο για αυτό το σημείο. Όχι, κανείς. Κύριε question. Ναι. Μια ερώτηση. Γιατί έχουμε καθυστερήσει. Είχε υποθεί αρχικά το πρώτο τρίμηνο για την εκπόνηση Είμαστε στον Απρίλη. Είχαμε και το Συμβούλιο πέρσι που είπε ότι αποτελεί μία από τις πιο επιτυχημένες πρωτοβουλίες και περιβαλλοντικά και, και οικονομικά κτλ. Οπότε τι γίνεται. Από ό,τι ξέρω και η Κομισιόν θέλει να ενισχύσει την αποτελεσματικότητα μέσω του σχεδίου για την κυκλική οικονομία. Υπάρχουν λοιπόν όλοι οι όροι και προϋποθέσεις, αλλά δεν προχωράει και αυτό δημιουργεί ανασφάλεια. Δεν καταλαβαίνω λοιπόν γιατί υπάρχει αυτή η μεγάλη καθυστέρηση τη στιγμή που έχετε σήματα από το Κοινοβούλιο, από το Συμβούλιο, από τη Βιομηχανία, από τη ΣΜΙΟ κτλ. ότι ενδιαφέρονται. Τι σας καθυστέρει, τι προκαλεί την καθυστέρηση, μπορείτε να μας πείτε κάτι παραπάνω. Γιατί αρχίζουμε πραγματικά να ενοχλούμαστε από την καθυστέρηση αυτή σήμερα. Ευχαριστώ κύριε Σπεντιτσίνη. Ναι, πρόεδρε, ευχαριστώ. Με ενδιαφέρον ακούσαμε εμείς την τοποθέτηση της Κομισιόν για το έμας και την οικοσήμανση. Αλλά πραγματικά χωρίς μελέτη αντικτύπου δεν μπορούμε να αποτιμήσουμε και να αξιολογήσουμε τις επιπτώσεις αυτών των πρωτοβουλειών. Η Επιτροπή μας όμως είναι υπέρ οποιασδήποτε πρωτοβουλίας που αφορά του καταναλωτές και που μειώνει τον κύκλο ζωής και τις επιπτώσεις των περιβάλλων προϊόντων. Με τρόπο ώστε να βοηθήσουμε και τις επιχειρήσεις να φανούν περισσότερο στην αγορά και να είναι πιο ανταγωνιστικές. Πάντως, για το αίμα και την οικοσήμανση θα πρέπει να προσέχουμε κατά πόσο θα καθοδηγήσουμε τους καταναλωτές σε συγκεκριμένε επιλογές για να μην δημιουργήσουμε σύγχυση σε σχέση με άλλες πληροφορίες οι οποίες περιλαμβάνονται στη σήμανση. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ανταλή. Ευχαριστώ πρόεδρε. Έχω την εντύπωση καμιά φορά ότι είναι ένας φαυλός κύκλος. Δηλαδή με την καθυστέρηση προκαλούμε υποχώρηση ενδιαφέροντο από ό,τι κατάλαβα από την παρουσίαση τη Κομισιόν. Εντάξει, υπάρχουν καθυστερήσει στην πρόσληψη, το κατανοώ αυτό. Κατανοώ επίση ότι δεν έχουμε αξιολογήσει πλήρω τον αντίκτυπο, αλλά όσο πιο καθυστερούμε, τόσο πιο σοβαρά θα είναι τα εμπόδια. Οπότε συμφωνώ με αυτά που άκουσα να υπάρχει δηλαδή κάτι το παραδοτέο, το οποίο επιτέλου θα παραδοθεί και να μην χρειάζεται να περιμένουμε άλλο. Πρέπει και η Κομισιόν να δει πώς θα το κάνει πιο ευπαρουσίαστο αυτό, πιο δημοφιλές. Θα ήταν λοιπόν καλό και εμείς να κατανοήσουμε και να δούμε περισσότερη διαφάνεια για το πώς εσείς προσπαθείτε να το αντιμετωπίσετε αυτό. Έστω και στις αρχικές φάσεις. Δηλαδή, σε ποιους τομείς θέλετε να επικεντρωθείτε και ποια κατεύθυνση θέλετε να ακολουθήσετε, ώστε και εμείς τέλο πάντων σαν Κοινοβούλιο να έχουμε μια ιδέα για το πού θέλει να πάει η Κομισιόν, έστω και στις πρώιμες φάσεις και να συνοδεύσουμε και εμείς την Κομισιόν στις προσπαθίες της. Ευχαριστώ κύριε Κονέσκα. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Πρόεδρε. Συνάδελφοι, θα ήθελα να προσθέσω κάτι σε αυτά που είπαν και οι συνάδελφοι. Δεν καταλαβαίνω γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αντιστέκεται σε κάτι το οποίο τη ζητά και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τα κράτη-μέλη. Στο Συμβούλιο έχει συζητηθεί αυτό το θέμα και η πλειοψηφία των κρατών μελών είπαν ότι θα έπρεπε να δράσει διαφορετικά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είναι κάπως απομονωμένη λοιπόν στο πρόβλημα αυτό η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο. Όλη την ώρα λέμε ότι ε, η οικοσήμανση είναι ένα ε, εργαλείο το οποίο βοηθά ε, τη δεσμευτική νομοθεσία και μπορεί να ενισχύσει την προστασία των περιβάλλοντος μέσω της αλλαγής συμπεριφοράς των καταναλωτών. Οι καταναλωτές το θέλουν, το κοινοβούλιο το θέλει, τα κράτη-μέλη το θέλουν αυτό που μας λείπει μόνο είναι η απόφαση. Και θα ήθελα να ξέρω για ποιο λόγο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, προχωρά κατά αυτόν τον τρόπο και μήπως θα μπορούσατε να μας δώσετε και επίσης ε, μια ημερομηνία γιατί το 2015 έγινε μια, ε, υπήρξε μια έκθεση, το 2016 έπρεπε να έχει γίνει μια αναθεώρηση, μια, αξιολόγηση, μια αξιολόγηση, η αξιολόγηση δεν έγινε το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ε, το συζήτησε και τώρα έχουμε μπει σε αυτό τον φαύλο κύκλο, όλοι το θέλουν, όλοι το ζητούν, όλοι το συζητούν, αλλά τελικά δεν υπάρχει. Μπορείτε να μας δώσετε μια, ένα ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα, όχι μια υπόσχεση απλώς. So, uh, Λοιπόν, Ευρωπαϊκή Επιτροπή για το συμπέρασμα. Λοιπόν, ναι, ε, λίγο περισσότερο χρόνο μας πήρε από ό,τι περιμέναμε, αλλά είμαστε στα τελικά στάδια. Στα τελικά στάδια είμαστε ε, για, τα πολιτικά συμπεράσματα του τι θέλουμε να κάνουμε με αυτά τα δύο μέσα και ελπίζουμε ότι ο πολιτικός προσανατολισμός... Ε, ε, του ε, σώματος των επιτρόπων θα ολοκληρωθεί σύντομα. Είναι γεγονός ότι το Συμβούλιο μας είπε ότι τα μέσα είναι επιτυχή, αλλά ε, αυτό πρέπει να το δείτε με λίγη προσοχή. Γιατί αν οι υπουργοί μίλησαν θετικά για αυτά τα δύο μέσα, για ποιο λόγο έχουμε τόσο χαμηλό επίπεδο καταχώρησης του ΕΜΑΣ, και τόσο λίγα προϊόντα με οικοσήμανση, αν είναι τόσο επιτυχημένο αυτό το, το μέσο. Την ερώτηση αυτή την κάνω και για τον εαυτό μου, αλλά πρέπει να αναρωτηθούμε πραγματικά 20 εκατομμύρια εταιρείες έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μόνο 4.000 καταχωρήσεις του ήμας. Ε, πώς γίνεται αυτό. Μπορούμε να το θεωρήσουμε αυτό επιτυχία δεν είμαι πολύ βέβαιος. Για να μπορέσουμε να το αποκαλέσουμε επιτυχία, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι τουλάχιστον 20% ε, των εταιριών, των ε, προϊόντων με τις καλύτερες επιδόσεις, ε, χρησιμοποιούν ένα από τα δύο προγράμματα. Τότε θα το αποκαλέσω ευχαρίστως επιτυχία. Α είμαστε λοιπόν πολύ ειλικρινεί σε σχέση με το τι συμβαίνει, για ποιο λόγο δεν πήγαν τα πράγματα όπως θέλαμε ακριβώ και με ποιο τρόπο μπορούμε να προωθήσουμε το σήμα καλύτερα. Πράγματι, Έχουμε μια έκθεση που θα προκύψει από την αξιολόγηση της αποδοτικότητας. Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσουμε το πρόγραμμα μας ως εργαλείο ε, ρυθμιστικής ανακούφισης για τις εταιρείες. Δηλαδή αν κάποιος θέλει να ακολουθήσει αυτό το πρόγραμμα πρέπει να ακολουθήσει αυστηρές περιβαλλοντικές προδιαγραφές, ε, ε, κάποιος το επαληθεύει και κάποιος σου δίνει το σήμα κατόπιν αξιολόγησης της έκθεσης. Αν το κάνει κανείς αυτό μπορεί τότε να εξαιρείται από άλλες περιβαλλοντικές εκθέσεις και αυτό είναι ένα κίνητρο για τις εταιρείες να χρησιμοποιήσουν χρησιμοποιούν το σήμα ήμας Έχουμε παραδείγματα κρατών μελών που το κάνουν αυτό, αυτό λίγα, λίγα, αλλά το κάνουν. Και ε, όταν γίνεται αυτό υπάρχουν ε, έγγραφες. Κάποιες περιφέρειες ενδεχομένως το κάνουν σε μερικά κρατημέλη, αλλά δουλεύει όταν το κάνουν. Θα ήθελα λοιπόν ε, να πω ότι αυτό το παράδειγμα υπάρχει και θα ήθελα να το ε, αντιγράψω και σε άλλες περιοχές για να μπορέσουμε να αυξήσουμε τον αριθμό των εγγραφών που είναι κάτι το οποίο θα είναι υποφελέ και για τις εταιρείε και για το περιβάλλον αυτό όμω δεν είναι πανάκια. Υπάρχουν τα μέσα, υπάρχουν κανονισμοί, πρέπει να τους επιβάλλουμε, υπάρχουν κριτήρια για τα προϊόντα, έχουμε ε, κάποια κριτήρια ε, για το έμας αν ε, οι εταιρείε, ο δημόσιος τομέας θέλει να τα χρησιμοποιήσει θέλουμε προώθηση ε, και δεν θέλουμε να παρεμποδίζονται οι εταιρείε από το να χρησιμοποιούν αυτό το σήμα. Θέλουμε να κάνουμε αυτόν τον έλεγχο αποδοτικότητας ε, του, κανονιστικού πλαισίου για να δούμε πώς μπορούμε να ε, αντιμετωπίσουμε κάποια προβλήματα. Όσον αφορά τον, την πληροφόρηση που ε, αφορά το συγκεκριμένο σήμα. Αυτό ενδεχομένω να είναι ένα πρόβλημα που πρέπει να λυθεί. Ε, ενδεχομένως το πρόβλημα είναι η πληθώρα των σημάτων και όχι τόσο η ενημέρωση για τα συγκεκριμένα προϊόντα. Αυτό είναι που δημιουργεί σύγχυση στους καταναλωτές. Μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν 500 με 1000 σήματα, πράσινα σήματα που δεν έχουν πάντοτε επαληθευτεί, δεν ελέγχονται από τις αρχές και αυτό είναι αυτό που πραγματικά δημιουργεί σύγχυση ε, στους καταναλωτές και καταστρέφει την εμπιστοσύνη τους. Πιστεύουμε ότι με αυτή την οικοσήμανση μπορούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα, αλλά μπορούμε να το λύσουμε μόνο αν είναι πολλές οι εγγραφές και αν καλύπτει πολλά προϊόντα και όχι μερικά μόνο προϊόντα. Για την ώρα 39.000 ε, προϊόντα με οικοσήμανση έχουμε από πάνω από ένα εκατομμύριο, μεταξύ πάνω από ε, ε, ε, ε ένα εκατομμύριο προϊόντα. Ε, πρέπει λοιπόν να βρούμε τη λύση σε αυτό. Γι' αυτό καθυστερούμε λίγο περισσότερο από ό,τι αναμενόταν και θέλουμε να πετύχουμε. Γιατί πρόκειται για κάτι που έχει τεράστιο δυναμικό. Αυτά τα σήματα πρέπει να προωθηθούν με το σωστό τρόπο και αν χρησιμοποιούνται βέβαια για καλούς σκοπούς, η κυκλική οικονομία είναι ένας καλός σκοπός ε, για τη χρήση τους. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει Πρόεδρος. Το τελευταίο σημείο στην, στην ημερήσια διάταξή μας ανταλλαγή απόψεων με το ECDC, το Ευρωπαϊκό Κέντρο για την ε, πρόληψη και την, ασφα... για την ε, πρόληψη και τον έλεγχο των ασθενειών. Σε σχέση με το ΖΙΚΑ. Η κυρία Λεμόν. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι εδώ σήμερα και μπορώ να σας παρουσιάσω τη δουλειά που κάνουμε για τον ΖΙΚΑ. Η ζήκα δεν είναι καινούρια αρρώστια. Την παρακολουθεί το κέντρο μας από το 2009, από όταν ξεκίνησε στην Αμερικανική Ήπειρο το 2015, το παρακολουθούμε στενά. Και ειδικά από τον Νοέμβριο του 2015, όταν το Υπουργείο Υγείας Βραζιλίας είπε πως υπάρχει κίνδυνος για τη δημόσια υγεία καθώς υπάρχουν, υπήρχε αύξηση στον αριθμό παιδιών που γεννιόνταν με μικροκεφαλία. Επίσης στη γαλλική Πολυνησία αναφέρθηκε μια εκ των υστέρων αύξηση συγγενών ανομαλιών ε, στα παιδιά το 2014 και 2015 που συνέπεσε με το πρώτο ξέσπασμα του ιού στο αρχιπέλαγο. Σε αντίδραση κάναμε μια γρήγορη αξιολόγηση κινδύνου το Δεκέμβριο 2014 και ακριβώ αναφερθήκαμε στην αύξηση των περιπτώσεων αυτών με νευρολογικές επιπτώσεις στη Γαλλική Πολυνικία και ακολούθησε μετά μια αξιολόγηση της επιδημίας και την πιθανή σχέση με την μικροκεφαλία. Την 1η Φεβρουαρίου του 16 ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας μίλησε για κατάσταση αναγκής διεθνούς ε, ενδιαφέροντος ε, που αφορούσε τα κρούσματα μικροκεφαλίας στις περιοχές που είχαν τον ιό και αύξησε το επίπεδο συναγερμού για να ανταποκριθεί δε η Κομισιόν, ε, τα κράτη-μέλη και τα ΜΜΕ φροντίσαμε να ανοίξουμε κάποιες γραμμές επικοινωνίας, όπως επίσης και με διεθνείς εταίρους μας, όπως τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, τον Παναμερικανικό Οργανισμό Υγείας, το ΤΑΧΟ, και βεβαίως ε, με τα κράτη-μέλη του ε, ΕΟΧ. Και βεβαίως ε, είχαμε το κέντρο επιχειρήσεων για να έχουμε ενιαία μηνύματα προς τα έξω. Κάναμε λοιπόν μία αναθεώρηση των σχεδίων ανάγκης για τις αρρώστιες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών για να ενισχυθεί επίσης η διεπιστημονική συνεργασία, να εμπλακούν οι κοινότητες ακριβώς για τους φορείς, τα κουνούπια φορείς ε, του Ιουζίκα και επίσης να δούμε και το τι γίνεται με τα χώροκαρακτητικά είδη. Κατόπιν ο ΠΟΕ στις 18 Νοέμβριο πέρσι είπε ότι έληξε πλέον η κατάσταση διεθνούς συναγερμού. Παρ' όλα αυτά εμείς συνεχούμε να παρακολουθούμε στενά την κατάσταση και εκδίδουμε και ταξιδιωτικές οδηγίες για τις πληγήσεις χώρες. Μέχρι στιγμής είχαμε 10 γρήγορες αξιολογήσεις κινδύνου. Η πιο πρόσφατη ήταν στις 10 Απριλίου πριν από λίγες εβδομάδες και 42 επιδημιολογικές ενημερώσεις. Αυτό αποδεικνύει πως ε, παρά το ότι η εντολή μας είναι να λειτουργούμε εντός των συνόρων της Ένωσης, οι απειλές από μεταδοτικές ασθένειες που εμφανίζονται οπουδήποτε στον κόσμο μπορούν να έρθουν στην Ευρώπη. Επίσης, δείχνει την σημασία της ευρωπαϊκής και διεθνούς συνεργασίας. Θα δώσω τώρα τον λόγο στην συνάδελφο Αβιτσέλερ, που είναι επικεφαλής ε, του προγράμματος μεταδοτικών ασθενειών στο ECDC, ο οποίος σας ενημερώσει για την επιδημιολογική κατάσταση και τον πιθανό κίνδυνο για την Ευρώπη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνετε αυτή την ενημέρωση εγώ θα έλεγα ότι αυτή η νόσος, η ασθένεια του Ζήκα είναι κάτι το οποίο υπήρχε στην Ασία, στην Αφρική, στο παρελθόν, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις ε, ήταν μία ασθένεια ε, εξανθηματική με πυρετό ε, και συνήθως η λοιμώδης νόση έτσι είναι, δεν έχουν συμπτώματα ε, που σημαίνει ότι μπορεί να υπάρξει και κύκλος μετάδοσης της νόσου από τα κουνούπια. Αλλά αυτό που συνέβη στη Γαλλική Πολυνησία και μετά στην βορειοανατολική Βραζιλία στην αρχή και μετά σε όλη την Αμερικανική Ήπειρο ήταν ε, ε, κάτι το οποίο εντοπίστηκε το 2015, όμως ε, δεν έχει σχέση με το σύνδρομο Γιγέν Βαρών, το οποίο αναφέρθηκε πρώτη φορά το 2013-2014 στη Γαλλική Πολυνησία και μετά στην, σε ολόκληρη την Αμερικανική Ήπειρο. Ε, και στην Ασία υπήρξαν ε, κάποια κρούσματα που αναφέρθηκαν. Ε, η μεγάλη απειλή ήταν αυτά τα συναφή σύνδρομα, συγγενή σύνδρομα, τα οποία εμφανίστηκαν στην Βραζιλία το 2015, σε κάποια μέρη της Βραζιλίας. Εκεί υπήρχε τεράστια ανησυχία ε, που είχε ως αποτέλεσμα αυτήν την ε, κατάσταση εκτάστου, ε, εκτάκτου ανάγκης και αν, αντικατα, αν, υποχρεωθήκαμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις απειλές. Ε, όταν υπάρχει μια επιδημία του ΖΙΚΑ υπάρχει περίπτωση να υπάρχει 30% αυξημένος κίνδυνος ε, γεννήσεων βρεφών με μικροκεφαλία ή με συγγενή προβλήματα του νευρικού συστήματος. Ε, υπάρχουν πάντως σοβαρές προκλήσεις ε, γιατί είναι μία ήπιας μορφής ασθένεια στον άνθρωπο μπορεί να γίνει εργαστηριακά η διάγνωση και η επιβεβαιώση της ασθένειας. Μία ανησυχία είναι ότι μπορεί να μεταδοθούν ε, και μέσω σεξουαλικής επαφής αυτές οι ασθένειες. Ε, υπήρχε μία τέτοια περίπτωση το 2011 και μετά κάποια ακόμη κρούσματα πιο μετά στην Ευρώπη ε, και στην Αμερικανική Ήπειρο και αυτά όλα εμφανίστηκαν εντός τριών εβδομάδων από τη μόλυνση ε, του άνδρα ε, τρεις εβδομάδες μετά. Εμφανίστηκε ε, μέσω σεξουαλικής επαφής στη γυναίκα. Τρεις εβδομάδες λοιπόν μετά από την εμφάνιση των συμπτωμάτων, αλλά επίσης υπάρχει και εντοπισμό στο γονιδίωμα και μετά από έξι μήνες. Τι σημαίνει αυτό, σημαίνει ότι υπάρχει κίνδυνος ε, ε, σεξουαλικής, ε, μετάδοση με σεξουαλική επαφή και έξι μήνες μετά εφόσον ανοιχνεύεται ακόμη ο ιός. Το πιο προληπτικό μέσο λοιπόν μέτρο σε σχέση με τις νέες αυτές απειλές ήταν η προστασία των εγγύων γυναικών, των γυναικών που θέλουν να συλλάβουν ε, και των ε, ε, εμβρίων. Έπρεπε λοιπόν να γίνεται, να υπάρχει ασφαλή σεξουαλική επαφή. Αυτό ήταν το περιοριστικό μέτρο το οποίο προτάθηκε έξι μήνες για τους άντρες και οχτώ εβδομάδες για τις γυναίκες στην Ευρώπη. Και αυτό συνάδει βέβαια με αυτό που προτάθηκε στην Αμερική και στη Βραζιλία. Όσον αφορά τώρα την επιδημιολογία και ο Ζήκα μειώνεται. Αν δείτε ας πούμε τι γίνεται στην Κολομβία, από ε, την 1η Ιανουαρίου μόνο 300 ε, ύποπτες ε, ε περιπτώσεις ε, έχουμε εντοπίσει και αν δούμε για παράδειγμα την Καραϊβική, Μαρτινίκα και Γουαδελούπη δεν έχουμε ε, καινούργια κρούσματα κατά, τελευταίους, κατά τους τελευταίους τρεις μήνες. Στην Αργεντινή μόνο μερικέ, μερικά κρούσματα το Φεβρουάριο. Ε, κάποια σποραδικά κρούσματα στην Αγγόλα, Σιγκαπούρη, Ταϊλάνδη, Φιλιππίνες και στον Ειρηνικό ωκεανό κανένα κρούσμα προσφάτως. Ε, Δεν ξέρουμε βέβαια τι θα γίνει, πρέπει να επαχρυπνούμε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει όταν θα αρχίσουν να εμφανίζονται και πάλι τα κουνούπια στην Αμερικανική Ήπειρο και στην Καραϊβική. Δεν θα, υπήρξε, δεν θα υπάρξει βέβαια επιδημία παρόμοια με τις περασμένες χρονιάς. Και για την Ευρώπη ε, ζητήσαμε από τα κράτη-μέλη να αναφέρουν ε, τους ε, ταξιδιώτες που έρχονται από περιοχές μολυσμένες για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε κατά πόσο υπάρχει κίνδυνος ε, εξάπλωσης του ιού στην Ευρώπη. Το 2016 βλέπουμε εδώ έναν χάρτη ενός από τους φορείς που μπορεί να μεταφέρει τον ιό, δηλαδή το μοσκίτο, το κουνούπι έντες αλμπόπικτους, ε, υπάρχει βέβαια και εξάπλωση και σε άλλες περιοχές. Πέρσι υπήρχαν 2.000 κρούσματα που αναφέρθηκαν και 1.000 εξ αυτών αναφέρθηκαν σε περιοχές όπου υπήρχε αυτό το κουνούπι. 30% ε, από τον Ιούλιο μέχρι τον Αύγουστο όταν είναι πολύ ενεργό αυτό το κουνούπι. Ε, υπάρχει λοιπόν μια πιθανότητα ε, επανεμφάνισης, υπάρχουν καλές κλιματικές συνθήκες για εξάπλωση ε, τοπικά του ε, ιού Ζήκα. Να δούμε τώρα ε, τι γίνεται με τους ταξιδιώτες. Ε, ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείου, προ, Υγείας προτείνει μία ταξινόμηση ε, αναζώνη, μία κατηγοριοποίηση, περιοχές με πρόσφατα ακρούσματα από το 2015 όταν έφτασε στις Αμερικανικές Υπήρους ο ιός, ε, ε, περιοχές στις οποίες υπάρχει ε, προηγούμενη αναφορά κρουσμάτων ε, και οι περιοχές με το γκρι που είναι περιοχές στις οποίες ενδεχομένως να εξαπλωθεί ο ιός αλλά δεν έχουμε πληροφορίες γύρω από αυτό και με το ανοιχτό γκρι είναι ε, οι περιοχές, το, οι περιοχές οποίες το κουνούπι που είναι υπεύθυνο και για το δάγκιο πυρετό, το έντες αλμπόπικτους, το έντους Αιγύπτη, ε, έχουμε λοιπόν για όλες αυτές τις περιοχές και κάποιες, κάποιους χάρτες ε, περιοχών που παρουσιάζουν αυτήν την ταξινόμηση των χωρών και βλέπετε για παράδειγμα για την Ασία έχουμε μόνο σποραδικά ε, κρούσματα, αλλά ήταν περιοχές οποίες υπήρχε ήδη ο ιός και στην Καραϊβική για παράδειγμα ε, και εκεί μπορεί να υπάρχουν κάποιες περιοχές. Για να δούμε τώρα τι γίνεται, τι γίνεται με τα ε, μέτρα, τα προληπτικά και τα μέτρα ελέγχου. Τι μπορούμε να κάνουμε δεν υπάρχει θεραπεία για τον ιό, δεν υπάρχει δυνατότητα πρόληψης της ε, μετάδοσης του ιού από τον πλακούντα στο έμβριο ε, μπορούμε να έχουμε λοιπόν μεμονωμένα προληπτικά μέτρα που είναι τα εντομοαποθετικά, η σωστή ένδυση, αλλά καταλαβαίνετε πόσο δύσκολο είναι αυτό να γίνει ε, η σωστή ένδυση, για παράδειγμα, σε τροπικές περιοχές και επίσης πρόληψη της μετάδοσης διασεξουαλικής οδού, ασφαλής λοιπόν σεξουαλική επαφή για τα ζευγάρια που θέλουν να συλλάβουν. Εν πάση περιπτώσει είναι κάτι το οποίο δεν μπορεί να είναι μακροχρόνια βιώσιμο ως ε, τακτική. Πρέπει να αντιμετωπίσουμε και τα κουνούπια, τα κουνούπια αλμπόπικτους και Αιγύπτιοι είναι παρόντα σε πολλές περιοχές, ε, τα βιοκτώνα δεν τους κάνουν τίποτα, δεν είναι ένα κουνούπι που είναι εύκολο να το ελέγξει κανείς, μπορεί να γίνει με τη χρήση ε, βιοκτώνων, κυρίως στους ενήλικους πληθυσμούς, αλλά και στα και στις προνύμφες, αλλά ε, πρέπει να προσπαθήσουμε να ε, είμαστε αποτελεσματικοί κυρίως στα σημεία παραγωγής των, των αυγοπαραγωγής των συγκεκριμένων κουνουπιών. Ε, Περιμένουμε ένα εμβόλιο για το 2020. Έχουμε ένα χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή Ένωση πρόγραμμα ε, για το ΖΙΚ, αλλά υπάρχει μια καθυστέρηση γιατί αυτό το ερευνητικό πρόγραμμα καθυστέρησε πάρα πολύ και έτσι αργήσαμε να αρχίσουμε. Ε, αρχίσαμε μόνο στο τέλος της ε, μεγάλης επιδημίας Υπάρχει λοιπόν ένα πρόβλημα με το χρονοδιάγραμμα, το οποίο πρέπει να το αναθεωρήσουμε για τέτοιου είδους επίγουσες καταστάσεις. Συμπερασματικά λοιπόν θα έλεγα ότι είναι μια ασθενής, ε, μια ήπια ασθένεια αυτή. Ε, πρέπει να υπάρξει διεθνής έλεγχος. Είναι μια ασθένεια που είπα ότι μεταδίδεται από τα κουνούπια Αλμπόπικτους και Αιγύπτη. Αυτό είναι ένα μια τεράστια ανησυχία. Ε, πρέπει να ελεγχθεί ο πληθυσμός αυτών των κουνουπιών. Είναι το πιο αποτελεσματικό μέσο. Είναι λοιπόν σημαντικό το συντομότερο δυνατό να κατανοήσουμε τη σημασία της ασθένειας και να έχουμε τα απαραίτητα εργαλεία για να μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε αυτούς τους παθογόνους παράγοντες και καλύτερη συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, μεταξύ των ε, διεθνών ε, υπηρεσιών, για να μπορέσουμε να αξιολογήσουμε την κατάσταση με τον καλύτερο τρόπο και εγκαίρως. Χρειάζεται επίσης ιδιαίτερη αισθέση, όπως είπε και η Ανδρέα Λεμόν προηγουμένως, να επικεντρωθούμε στην εποπτεία και στην, ε, στο να είμαστε έτοιμοι, στην ετοιμότητα. Ευχαριστώ πολύ. Δίνω το λόγο τώρα στην κυρία Κονέτσνα, που είναι το, η συνάδελφος επαφής μας. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Να ευχαριστήσω αυτή την υπηρεσία για τα θαυμάσια δουλειά της στον τομέα αυτό. Πιστεύω ότι μέσω της τεχνογνωσίας και της ανταπόκρισης, όχι μόνο για το ΖΙΚΑ και το ΕΠΟΛΑ, αλλά και για άλλα θέματα, έχει αποδείξει την ανάγκη της υπαρξής της η υπηρεσία αυτή. Νομίζω ότι η συνεργασία μεταξύ των διαφόρων αντίστοιχων υπηρεσιών στις ε, χώρες της Ένωσης υπό την αιγίδα του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας θα πρέπει να ενισχυθεί και το ECDC θα πρέπει να παραμείνει ένα οργανισμός πρώτης γραμμής. Νομίζω ότι ο εμβολιασμό θα αποτελέσει λύση κλειδί στο μέλλον για την αντιμετώπιση αυτών των επιδημιών και μέσω ανάπτυξης του εμβολιασμού αυτού μπορούμε να προστατεύσουμε τους αυτούς μας από αυτούς τους κινδύνους που μπορεί να είναι και θανατηφόροι όπως στην περίπτωση του έμπολα. Επειδή είδαμε και σε περιπτώσει άλλων πρόσφατων ασθενειών την ανάπτυξη, δυνατότητα ανάπτυξη εμβολιασμού και ελπίζουμε να συμβεί και εδώ κάτι, τέτοιο. Ελπίζω βέβαια και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να υποστηρίξει το ECDC για το θέμα αυτό, γιατί πραγματικά μπορεί να μας επηρεάσει στην Ευρώπη, αλλά έχουμε εμπειρογνώμονες, έχουμε αρχές, έχουμε τεχνογνωσία ώστε να αντιμετωπίσουμε αυτούς τους κινδύνους. Βέβαια, δεν θα θέλαμε να βλέπουμε να επαναλαμβάνεται αυτή η κατάσταση, αλλά είναι καλό γενικά να ξέρουμε ότι υπάρχει ένας αξιόπιστος οργανισμός αντιμετώπισης και το ECDC νομίζω πράγματι απέδειξε τη χρησιμότητά του και να ευχαριστήσω όλους τους εμπλεκόμενους, όλους τους υπαλλήλους του οργανισμού για την καταπολέμηση αυτών των επιδημιών και των ασθενειών. Νομίζω ότι πραγματικά βοηθήσατε όλες τις χώρες μέλη να αντιμετωπίσουν καλύτερα τα φαινόμενα αυτά. Ίσως θα πρέπει να βρούμε και ένα ταχύτερο μηχανισμό που θα επιτρέπουν μεγαλύτερη ανταπόκριση αλλά ευχαριστώ και πάλι πολύ την ECDC για όλη τη δουλειά που έχει κάνει. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ντόναν. η κυρία, συγγνώμη, Ντονανό. Ευχαριστώ το ECDC, λέει κύριε Ντονανό για την παρουσίαση σχετικά με το ΖΙΚΑ. Ο κίνδυνος στην Ευρώπη δεν είναι μελητός όχι μόνο των μετακινήσεων στις ζώνες κινδύνου, αλλά και ε, λόγω των υπερπόντων ενταφών. Ο Παγκόσμιο Οργανισμό Υγεία έχει ταξινομήσει την Γαλλική Πολυνησία ω ε, περιοχή κινδύνου 3. Υπάρχουν όμω και άλλε περιοχέ όπω η Γουαδαλούπη, η Μαρτινίκη κτλ. όπου έχουμε οροθετικότητα δωρητών αίματος αρκετά υψηλή, κάτι το οποίο είναι ανησυχητικό. Σχετικά τώρα με την δωρεά οργάνων, σε αυτές τις ε, περιοχές προβλέπετε έναν προληπτικό έλεγχο αυτών των φαινομένων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Ανταλή. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Είχαμε πρόσφατα μια κινητοποίηση σε σχέση με τα κουνούπια, όπου οι επιστήμονες παρακολουθούσαν φαινόμενα που αφορούν τις ασθένειες που μεταδίδονται μέσω κουνουπιών, ώστε να κατανοήσουμε όλοι το πώς μετακινούνται αυτά τα είδη κουνουπιών, πώς μεταφέρουν τις ασθένειες, αλλά και ταυτόχρονα για να παράσχουμε πληροφορίες στους επαγγελματίες του μιας υγείας και στους πολίτες για να αντιμετωπίσουμε τους κινδύνους. Ήθελα λοιπόν να ρωτήσω το ECDC μήπως μπορούν να επιβεβαιώσουν ακριβώς σε ποια κατάσταση βρίσκεται αυτή η πρωτοβουλία για τα κουνούπια και ποιες είναι οι απόψεις τους σε σχέση με το κουνούπι τίγρη και τον ρόλο του στην εξάπλωση του ΖΙΚΑ. Θα μπορούσαμε λοιπόν να ενισχύσουμε προγράμματα ενημέρωσης των πολιτών ιδιαίτερα όσον αφορά την ύπαρξη και τη μετάδοση αυτών των ασθενειών από τα κουνούπια. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, λέει και πρόεδρος, ο κ. Χώσεν. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρουσίαση της κατάστασης, αλλά τώρα που έχει φύγει το θέμα από τα πρωτοσέλιδα, τι γίνεται, υπάρχει κάποια παύση ή δεν είναι τόσο πολλά τα κρούσματα. Ε, είπατε ότι εντάξει δεν είναι ακριβώς και ε, αυλαβής η ασθένεια, αλλά είπατε ότι δεν ξέρουμε και τι θα γίνει με την επόμενη εποχή των κουνουπιών. Υπάρχει κάποιο, ε, δεν ξέρω, κατώτατο επίπεδο ή θα υπάρξει κάποια αλλαγή ή δεν είναι τόσο μεγάλο το πρόβλημα ή δεν ξέρουμε τι θα γίνει τα επόμενα χρόνια. Έχουμε, θυμόμαστε ακόμα τις εικόνες που είχαμε δει από τη Βραζιλία όπου χρησιμοποιήθηκαν εντομοκτώνα για τα κουνούπια. Είπατε ότι δεν βοηθάει αυτό γιατί ήδη μεγάλα κομμάτια των κουνουπιών ε, τίγρεων είχαν αναπτύξει ανοχή στα βιοκτώνα. Οπότε δεν πρέπει να στηρίζουμε πια τέτοια μέτρα με βιοκτώνα. Γιατί έτσι αυξάνεται και ο κίνδυνος ε, αντοχής. Επίσης είπαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ότι θέλουμε να στηρίξουμε τις χώρες που πλήττονται περισσότερο τι έχει κάνει η Ευρωπαϊκή Ένωση. για να μπορέσουμε έτσι προσεχώς να ελέγξουμε την αρρωστία. Σας ευχαριστώ. Επανερχόμαστε στην κυρία Νομών για τις απαντήσεις. Σας ευχαριστώ. Θα ξεκινήσω με τις απαντήσεις και θα συνεχίσει ο συνάδελφος. Πρώτα απ' όλα, σας ευχαριστώ για την εκτίμηση που δείχνετε στην δουλειά μας. Είναι σημαντικό να θεωρείτε σημαντική την δουλειά μας και να χρησιμοποιείτε για δράσεις στις χώρες. Θα ήθελα να αναφερθώ στο θέμα τη σύσταση ε, ελέγχου της αιμοδοσίας. Ναι, βεβαίως κάτι τέτοιο το σύστημα, αλλά βεβαίως τα, τα πει και ο συνάδελφος αυτά. Για την στήριξη οργανισμών, ε, δυστυχώς, τέλος πάντων έχει δυστυχώς, εμείς ε, μπορούμε να δώσουμε στήριξη μόνο κατόπιν διαγωνισμού. Θα πρέπει λοιπόν να γίνει μια προκήρυξη. Δεν μπορούμε απευθείας να στηρίξουμε κάποιου οργανισμούς ε, παρά το ότι κάνουν χρήσιμη δουλειά. Ε, θα πρέπει λοιπόν να υπάρχει κάποια προκήρυξη όπως σας είπα. Θα δώσω τώρα τον λόγο συνάδελφο. σε σχέση με τις ουσίες ανθρώπινης προέλευσης. Κοιτάξτε, θα σας πω, υπάρχει μια ανησυχία ενδεχόμενης μετάδοσης του ιού από το αίμα και αυτό ήταν η περίπτωση στη Γαλλική Πολυνησία το 13 με 14 και εκεί ε, φύρμωσαν εμολυψίες, ε, είχαν ε, μια πολιτική επί του θέματος για ένα χρονικό διάστημα μετά την επιδημία. Αυτό εφαρμόστηκε επίσης και σε κάποια υπερπόντια, σε κάποια υπερπόντια εδάφη όπως τη Μαρτινίκα και τη Γουαδελούπη. Ε, κατά τη διάρκεια της επιδημίας. Ε, πρέπει να έχουμε όμως μια συντονισμένη πολιτική ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση και υπάρχει τώρα μια αναθεώρηση των κατευθυντηρίων γραμμών σε σχέση με το ΖΙΚΑ και τις σχετικές ασθένειες για έλεγχο βάση ε, της επιδημιολογικής κατάστασης. Δηλαδή εξατάτε από την επιδημιολογική εποπτεία κατά πόσο θα χρειαστεί ή όχι να γίνει έλεγχος, να γίνουν ε, ε, εξετάσεις. επόμενη ενημέρωση θα λάβει χώρα τον επόμενο μήνα. Όσον αφορά τώρα την συμμετοχή των πολιτών, όσον αφορά τα κουνούπια. Αυτό είναι κάτι το οποίο ελήφθη υπόψη να αποκοινούμε το ECDC. Έχουμε ένα δίκτυο δημόσιας ε, ε, παρακολούθησης των επιδημιών και των ζωονόσων, δηλαδή χαρτογράφηση της εξάπλωσης ε, και της χαρτογράφησης των διαφόρων φορέων, στην περίπτωση αυτή των κουνουπιών, για να ενισχύσουμε την αντιμετώπιση του ΖΙΚΑ σε περιοχές όπου είναι παρόν το κουνούπι αυτό. Τότε όταν έγινε η εφαρμογή δεν ξέραμε κατά πόσο το κουνούπι αυτό ήταν πολύ καλός φορέας του ΖΙΚΑ. Σύμφωνα με εργαστηριακές δοκιμές, τα οποία όμως τα λάβαμε τα στοιχεία κάπως καθυστερημένα, ε, δεν είναι πάρα πολύ καλός φορέας του ΖΙΚΑ, δηλαδή είναι πολύ χαμηλότερη η δυνατότητα, η πιθανότητα μετάδοσης μέσω αυτού του κουνουπιού ε, σε σχέση με αυτό που περιμέναμε. Ε, υπάρχει ένα δίκτυο εντομολόγων ε, και έτσι τα κράτη-μέλη ενημερώνονται για τις διάφορες πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται, όπως για παράδειγμα υπάρχει μια παγκόσμια συμμαχία κουνουπιών που έχει ένα τέτοιο πρόγραμμα. Ε, βλέπουν τώρα οι χρήστες μέσω αυτού του δικτύου ε, μπορούν να δουν κατά πόσο υπάρχει παρουσία ενός κουνουπιού ε, στην περιοχή τους ή όχι. Και είναι σημαντικό να μην γίνεται άπαξη διασταύρωση μέσω αυτού του δικτύου. Πρέπει συνεχώς να το κάνουμε αυτό, τακτικά, Και ένα μήνα μετά πρέπει να δούμε κατά πόσο υπάρχει παρουσία του κουνουπιού και γι' αυτό ακριβώς έχουμε και αυτούς τους χάρτες. Χρησιμοποιούμε τέτοιου είδους ε, λοιπόν ε, ε, πρωτοβουλίες, αλλά αυτό γίνεται μέσω διαφόρων δικτύων ενομολόγων δεν γίνεται σε επίπεδο ECDC. Κοιτάξτε, για την πλήρη εξάλληψη του ΖΙΚΑ. Ε, Υπάρχουν κάποιες, ε, κάποια κρούσματα ακόμη σε κάποιες κοινότητες της Βραζιλίας και σε κάποια μέρη της Αμερικανικής Υπήρου. Ξέρετε ότι υπάρχουν τα συγγενή προβλήματα του νευρικού συστήματος που προκαλεί ο Ζήκα στην Αφρική. Ε, είναι όμως πάρα πολύ περιορισμένου, ε, περιορισμένη η εμφάνιση του φαινομένου αυτού. Υπάρχει ένα συγκεκριμένο pattern ε, ε, μετάδοσης. Μπορεί να υπάρχουν δεκάδες, ε, δεκαετίες χωρίς να εμφανιστεί καθόλου. Σκεφτείτε για παράδειγμα τον κίτρινο πυρετό στην Βραζιλία που δεν είναι τόσο μακριά από το Ρίο Ντετζανέιρο που, σε περιοχές όχι πολύ μακριά από το Ρίο Ντετζανέιρο κάνουν ακόμη εμβολιασμούς. πρέπει λοιπόν να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί. Πρέπει να συνδυάσουμε την ε, εποπτεία των κουνουπιών, την επιδημιολογική εποπτεία για να μπορούμε να δίνουμε τη σωστή ενημέρωση ώστε μια χώρα να αντιμετωπίσει την επιδημία αυτή. Και όσον αφορά την αντοχή σε χημικά των ε, φορέων, αυτό είναι μια πραγματική ανησυχία. Πρέπει να δούμε εναλλακτικέ μεθόδους. Υπάρχουν κάποιες υπό αλλά χρειάζεται περισσότερη έρευνα ως προς αυτό. Και επίσης πρέπει να πούμε Πρέπει να δούμε στην επόμενη παγκόσμια συνέλευση υγείας ε, τι θα παρουσιαστεί. Υπάρχει ένα παγκόσμιο ε, ε, πρόγραμμα το οποίο θα παρουσιαστεί και θα δούμε πώς θα το υποστηρίξουν οι χώρες. Επίσης συνεργαζόμαστε με τον ΠΟΗ και με άλλους διεθνείς οργανισμούς ως προς αυτό και όσον αφορά τον εμβολιασμό υπάρχει μια πραγματική ανάγκη εμβολιασμού κυρίως προς τις νεαρές γυναίκες. Τις νεαρές γυναίκες η Ευρωπαϊκή Ένωση υποστήριξε μέσω ενός προγράμματος, ε, ενισχύει την προσπάθεια μιας εταιρείας για την ανάπτυξη εμβολίου. Ευχαριστώ. Thank Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ όλους για αυτή τη συζήτηση. Αυτό ήταν το τελευταίο σημείο στην ημερήσια. Θα τα ξαναπούμε στις 3 το απόγευμα. Ευχαριστώ πολύ.